αγαπητοί συνάδελφοι, ήλθε η ώρα μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε και το πρώτο σημείο στη μέση διάταξη <clears throat> είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΕΝΒΗ, κύριο Φάλκενμπεργκ, για τη δέσμη μέτρων για τα απόβλητα. Όπως ξέρετε αυτό είναι κομμάτι μιας μακράς ιστορίας σε σχέση με την δέσμη αυτή μέτρων. Και τώρα θα περάσω στα Ιταλικά. Γιατί θέλω να πω κάτι πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Με συγχωρείτε που περνάω στα Ιταλικά, αλλά μου απλουστεύει την έκφραση για την παρουσίαση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ιστορικό αυτής της δέσμης μέτρων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Γνωρίζουμε ποια ήταν ε, η πορεία όταν το Κοινοβούλιο ξεκίνησε να επεξεργάζεται αυτό το νομοθετικό πακέτο. Η ακρόαση που θα κάνουμε σήμερα είναι μέρος αυτής της πορείας. Θα ξέρετε όλοι σας ότι είχαμε πάρα πολλές ε, συζητήσεις με την Επιτροπή για το πακέτο αυτό, για αυτή την δέσμη μέτρων και αρκετές διαφωνίες. Εδώ θέλουμε και να συνεχίσουμε την μελέτη του θέματος και την επεξεργασία. Είμαστε, πιστεύουμε, σε ένα από τα πρωταρχικά στάδια της μελέτης του όλου θέματος ως Επιτροπή Περιβάλλοντος και γι' αυτό ε, ζητήσαμε πολύ έντονα και με όλα τα διαθέσιμα μέσα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο ε, προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών ζητήσαμε την διατήρηση του, του πακέτου αυτού. Το σημείο το είδαμε και στην ε, τελευταία ολομέλεια με ένα ψήφισμα που συνολικά δεν υπερψηφίστηκε. Όμως οι τροπολογίες που αφορούσαν το συγκεκριμένο πακέτο πέρασαν. Άρα στο Κοινοβούλιο υπάρχει βούληση και διάθεση να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Κατά τα άλλα, κατά τη διάρκεια του διαλόγου μας ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ολομέλεια για το πρόγραμμα εργασιών της, ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει πρόταση ακόμη πιο φιλόδοξη σε σχέση αυτό που ήδη θεωρούσαμε και εμείς φιλόδοξο και που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε. Εξού και πιστεύω ότι ο σημερινός διάλογος με τον κύριο Φάλκενμπεργκ πρωτίστως και μετά με την ακρόαση που θα έχουμε θα είναι ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία διαλόγου των θεσμικών οργάνων αλλά και για την εμβάθυνση των γνώσεών μας από το θέμα θα δούμε αν από τα στοιχεία του διαλόγου προκύψουν ενδεχομένω προτάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ακόμη πιο φιλόδοξη πρόταση από εκείνη που έκανε. Όμω, επαναλαμβάνουμε, όπω κάναμε ανέκαθεν ω Επιτροπή ΕΝΒΗ, θέλουμε να συζητηθεί αυτό το πακέτο, αυτή η δεσμή μέτρων και θέλουμε να ε, συζητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο και με το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο τοποθετήθηκαν και πολλοί υπουργοί προκειμένου να διατηρηθεί αυτή, αυτό το πακέτο. Η πλειοψηφία των Υπουργών Περιβάλλοντος έγραψαν ε, σε επίπεδο Συμβουλίου έγραψαν στην πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ώστε να διατηρηθεί το όλο πακέτο. Εν αναμονή λοιπόν της τελικής απόφασης από την πλευρά της Επιτροπής, προχωρούμε. Προχωρούμε με το σημαντικότατο αυτό ορόσημο στην όλη μας πορεία. Σε αυτή τη φάση να δώσω αρχικά το λόγο στο, στη συνάδελφη στον συνάδελφο Μποναθέ, στη συνάδελφο Μποναθέ για την αρχική της ε, παρουσίαση. Θα την παρακαλέσω να παραμείνει στα 5 λεπτά και μετά στον ε, Γενικό Διευθυντή Φάλκενμπεργκ. Παρακαλώ κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή Φάλκενμπεργκ για την παρουσία του μεταξύ μας. Όπως είπατε πρόεδρε, θα ήθελα να έχω κάνει μια παρέμβαση διαφορετική για να περάσω στην ουσία της όλης πρότασης, αυτού του σημαντικότατου ντοσχέ που εξετάζουμε. Διότι αναμφίβολα υπάρχουν κάποια σημεία ε, ισχυρά στην πρόταση ε, και κάποιες αδυναμίες. Για πρώτη φορά λόγω χάρη έχουμε μια μέθοδο υπολογισμού της ενιαίας ανακύκλωσης που συνδυάζεται με πιο φιλόδοξους στόχους και την απαγόρευση ως το 2030 να ε, μεταφέρονται απόβλητα στις χωματερές. Αυτό είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία της πρότασης όπου θα μπορούσαμε να ασκήσουμε επικριτικά σχόλια. Δηλαδή χρειάζεται περισσότερη μελέτη σε τα σημεία αυτά. Αυτό θέλαμε να κάνουμε σήμερα και ε, διατηθέμεθα να το κάνουμε και τις ερχόμενες εβδομάδες. Όμως για τους λόγους που αναφέρατε προηγουμένως και για όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, η συζήτηση τελικά στη σημαντική αυτή πρόταση μετατοπίστηκε από την ουσία στι στις φήμες. Εγώ θα προτιμούσα να μιλάω για παρασκήνιο, διότι σήμερα ακόμη πρόεδρε, το Κοινοβούλιο, εμείς δεν καταλάβαμε για ποιους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριλάβει την πρόταση αυτή μεταξύ όσων δεν θα εξεταστούν το 2015 στο πρόγραμμα εργασιών, δηλαδή αποσύρθηκε. Βέβαια, καλώς ε, πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να θυμίσω για το ιστορικό της πρότασης, για όσους δεν είναι μήμεροι, ότι υπήρξε ε, μια επιστολή ανάθεσης καθηκόντων του Πρόεδρου Γιούνκερ προς τον Επίτροπο Βέλλα, όπου ζητούσε να αξιολογηθεί η κατάσταση του όλου πακέτου βάσει των πρώτων αντιδράσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ότι έπρεπε να επανα υποτιμηθεί η συνοχή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σκοπούς ανάπτυξης και απασχόλησης. Έπειτα είχαμε ακρόαση, ακρόαση του Επιτρόπου Βέλα, όπου υπερασπίστηκε το πακέτο αυτό και ως πρώτη προτεραιότητα της θητείας του ανέφερε την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, στην οποία ανήκει και το πακέτο αυτό για τα απόβλητα, αλλά τελικώς που καταλήξαμε. Ο Αντιπρόεδρος, ο Επίτροπος Τίμερμανς, που ήρθε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου είπε ότι η πρόταση αποσύρεται. Και επίσης ότι θα υποβάλει εντός του 2015 νέα φιλοδοξότερη πρόταση. Και παραθέτω τα λόγια του, μια πρόταση που θα κλείνει τον κύκλο Καταλαβαίνω ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή είναι ως προς την ανάπτυξη της οικονομίας. Συμφωνώ και εγώ και μακάρι να πηγαίναμε και παραπέρα. Όμως το πρόβλημα είναι αυτό, ότι έχουμε και μια μελέτη αντικτύπου μπροστά μας. Τα γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Φάλκεμπερ, γιατί επ' αυτόν εργάστηκε και υπάρχουν και οικονομικά δεδομένα. 180 έως 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασιών λόγος σε αυτόν τον τομέα. Αύξηση του ΑΕΠ ε, κατά το 1% ακόμη και στο πλαίσιο της τεκλικής οικονομίας. Εξοικονόμηση πρώτων υλών. Μεταξύ του 10% και του 40%. Εάν λοιπόν ισχύει ότι θα έχουμε μια φιλοδοξότερη πρόταση ε, το ρωτώ και προς ε, τον κύριο Φάλκενμπεργκ. Τι θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο, να αυξηθούν ε, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, μακάρι. Σημαίνει ότι θα δούμε και άλλες διαστάσεις που δεν είναι μόνο αυτές των αποβλήτων. Και εκεί, μακάρι, αλλά τα όρια του 2015, διότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποβάλλει πρόταση εντός του έτους. Και στην περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, θα τηρήσετε την προθεσμία του 2015 ή θα καθυστερήσουμε κι άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, εάν εννοείται πιο φιλόδοξο να είναι πιο υψηλή στόχη. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να εργαστεί και από αύριο το πρωί, ιδίω αν μιλάμε για του στόχου τη πρόληψη. Αλλά γιατί να αποσυρθεί η πρόταση σε αυτή την περίπτωση και να μην αρχίσουμε ήδη από τώρα να εργαζόμαστε όλοι μαζί επί των νέων υψηλότερων στόχων. Συνολικά λοιπόν πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, κάποιες απορίες. Ε, όλοι, σε όλους μας γεννήθηκαν απορίες. Και κάτι ακόμα, πριν από έξι μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Άλλαξε βεβαίω η Επιτροπή, ε, είναι πολύ σαφέ το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε ένα συμβούλιο που εκφράστηκε ε, και είπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αποσύρει την πρόταση. Έχουμε μια πολύ ισχυρή έκφραση από πλευρά Κοινοβουλίου και το είδαμε στην τελευταία Ολομέλεια, όπου όντω δεν πέρασε κανένα ψήφισμα επί του προγράμματο, αλλά όπω το θυμήσατε κι εσεί, Πρόεδρε, Είχαμε ευρύτατη πλειοψηφία για τις τροπολογίες που ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αποσύρει την πρόταση. Και επειδή φαντάζομαι ότι εξήλυσα το χρόνο μου, δεν θα επαναλάβω τα λόγια ε, του Υπουργού Περιβάλλοντος, της Λετωνικής Προεδρίας που ακούσαμε χθες εδώ έχουμε πραγματικά μια υπαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οδεύω προς το τέλος. Είμαι φιλόδοξη ε, από χαρακτήρα. Έρχομαι από μια τέτοια χώρα και περιοχή. Γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταγράψει όλα τα σχόλια που θα ακούσει σήμερα και ελπίζουμε ότι θα ξαναδούμε τον, ε, τον διευθυντή Φάλκεμπερκ το Μάρτιο όταν θα ξανασυζητήσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Φάλκενμπεργκ για την ε, παρέμβασή του. Παρακαλώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την διοργάνωση αυτής της συνάντησης και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είναι γεγονός ότι όταν στις αρχές Δεκεμβρίου πήρα αυτή την πρόσκληση η εντύπωση μου ήταν λίγο σαν και αυτά που είπε η Σιμώνα Μποναφέ ότι θα συζητούσαμε τις λεπτομέρειες της πρότασης που είχε υποβάλει η Κομισιόν για τα θέματα αυτά, αλλά έκτοτε η νέα Επιτροπή αποφάσισε ότι η πρόταση αυτή δεν θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από την Κομισιόν με τη μορφή με την οποία είχε κατατεθεί. Αποφάσισε η Κομισιόν ότι θέλει να επανεξετάσει αυτή την πρόταση και να δει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μέσα από νομοθετικές πράξεις μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. και να συμβάλλει έτσι στην ε, δημιουργία ανάπτυξης που είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της Νέας Κομισιόν και που θέλει τόσο κατεπηγόντως να ξεκινήσει και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν και η Σιμώνα Βοναφέ το ανέφερε επίσης, έχει πάρει την απόφασή της, αλλά είπε συγχρόνως ότι θα επισημοποιηθεί αυτή η απόφαση αφού γίνει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εμεί έχουμε παρακολουθήσει πολύ κοντά, από πολύ κοντά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδαμε ότι δεν προέκυψε κάποιο ψήφισμα από το Κοινοβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό για το πρόγραμμα της Κομισιόν, το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Παρακολουθήσαμε όμως τη συζήτηση και έχουμε καταγράψει τις διάφορες αρκετά σαφείς απόψεις που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία και την καλύτερη αντιμετώπιση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και η οριστικοποίηση της πρότασης της απόφασης Κομισιόν αναμένεται να λάβει χώρα κάποια στιγμή στον Φεβρουάριο όταν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν περατώσει τις συζήτηση με την Κομισιόν. Μια πρώτη διευκρίνηση τώρα των ε, προθέσεων της Κομισιόν για την ε, απόσυρση αυτής της πρότασης. Η Κομισιόν έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταθέσει μια πληρέστερη και πιο φιλόδοξη πρόταση και αυτό θα γίνει μέσα στο ελεστός έτος, το 2015. Νομίζω και αυτό είναι μια σαφής ένδειξη του ότι η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στις συζητήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης συναρμόζεται με την Γενική Στρατηγική της Κομισιόν. Γιατί λοιπόν έχουμε μια νέα προσέγγιση. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα λεπτομεριακά πώς θα είναι η νέα πρόταση, γιατί είναι ακόμα υπό επεξεργασία. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η εκπόνηση της νέας αυτής πρότασης. Υπάρχουν όμως κάποιοι, κάποιες κατευθύνσεις, υπάρχουν κάποιοι τομείς αδυναμίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, που υπήρχαν στην παλιά πρόταση, κάτι το οποίο ακούσαμε και στις συζητήσεις με το Συμβούλιο, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος και φυσικά υπήρξαν πολλά σημεία τα οποία έχουν υποδειχθεί από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εξετάσει το θέμα της κυκλικής οικονομίας και έχουμε καταλήξει σε νομοθετικές προτάσεις που θα αντικαταστήσουν την τωρινή νομοθεσία πρόκειται για κάποια νομοθετικά στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως θα έπρεπε να τύχουν αναθεώρησης και η πρόταση που υπήρχε στο τραπέζι εστίαζε στην ε, αναθεώρηση αυτών των νομοθετικών μέτρων και έκανε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο φιλόδοξη και βελτία η νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επενδύσεις οι οποίες θα έπρεπε να εξευρεθούν και να υλοποιηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή η οποία θα υποστήριζε την ε, διαχείριση των αποβλήτων και όχι μονάχα πια την ε, πορεία προς τις χωματερές ενός μεγάλου μέρους από τα απόβλητα που παράγουν οι κοινωνίες μας. Είναι σαφές για μας όλους <clears throat> ότι κάθε χρόνο Υπάρχουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι που πηγαίνουν σε χωματερές, αποβλήτων πηγαίνουν σε χωματερές στην Ευρώπη, αυτό και κάθε χρόνο κιόλα, και επομένως πρέπει να βρεθεί μια καλύτερη λύση για αυτά τα προβλήματα. Στη νέα πρόταση, η Κομισιόν έχει αναφέρει το ότι θα ήθελε να εξετάσει το σύνολο της κυκλικής οικονομίας. Οι προτάσεις μας, οι νομοθετικές μας προτάσεις, αντιμετωπίζουν το τμήμα που έχει να κάνει με τα απόβλητα στην κυκλική αυτή οικονομία. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η ανακύκλωση θα πρέπει να απλοποιηθεί σημαντικά με την καλύτερη σχεδίαση των προϊόντων. Με την τροποποίηση του τρόπου που χρησιμοποιούμε κάποιες συγκεκριμένες ουσίες, ώστε να μπορούν να αποχωριστούν στο τέλος του, της ζωής του προϊόντος με το να λαμβάνουν υπόψη την τοξικότητά τους ώστε να αποφύγουμε προβλήματα όταν φτάνουμε στο στάδιο ανακύκλωσης αυτών των προϊόντων και έτσι ξέρουμε ότι για προϊόντα που έχουν τοξικές ουσίες είναι μεγάλη δυσκολία για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα υλικά δεύτερης γενιάς ή αλλιώς καταλήγουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε στο τέλος του κύκλου να ανακτήσουμε δευτερεύουσες ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να ανταγωνιζόνται πρωτογενείς πρώτες ύλες. Και αυτό είναι ένα στόχος τον οποίο όλοι θέλουμε να επιζητήσουμε. Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας προκύπτει από μια ανάλυση αποδοτικότητας των βασικών πόρων που δείχνει ότι αρχίζουμε να αντιμετωπίσουμε <clears throat> την περατότητα του πλανήτη μας και τα όρια των φυσικών πόρων, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής μας, αν θέλουμε να υπάρξει και έξοδος πολλών εκατομμυρίων στον αναπτυσσόμενο κόσμο από την τωρινή του ένδια, είναι απαραίτητο να έχουμε μια καλύτερη χρήση πρώτων υλών, καλύτερη αξιολόγηση των αποβλήτων, καλύτερη χρήση του φυσικού μας κεφαλαίου. Αυτός είναι ο στόχος που επιζητούμε να <clears throat> εξυπηρετήσουμε και αυτό που θέλει να προωθήσει η Κομισιόν είναι μια αναθεωρημένη πρόταση η οποία θα συμπεριλάβει όλα τα διδάγματα της καλύτερης ρύθμισης, θα λάβει υπόψη τις ερωτήματα επικουρικότητος για το πώς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε με το βέλτιστο τρόπο να προχωρήσουμε, να εξασφαλίσουμε ότι απλώς δεν αποφασίζουμε να περάσουμε νομοθεσία και μόνο, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως, μια αντιμετώπιση που λαμβάνει υπόψη και τις επενδυτικές ανάγκες. Και όταν αρχίζουμε λοιπόν την επανεξέταση εν ώψη της τροποποίησης των προτάσεων που είχε υποβάλει η Επιτροπή Μπαρόζο. Εμείς ήδη συμπεριλαμβάνουμε ορισμένα σχέδια δημιουργίας περιβαλλοντικής υποδομής στα σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να τύχουν χρηματοδότησης από το λεγόμενο ε, σχέδιο επενδύσεων ή την πρωτοβουλία επενδύσεων Juncker. Έχουμε λοιπόν καταλήξει ορισμένε ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μοχλεύσουμε σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων. Εξετάζουμε τους τομείς και τα σχέδια που θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποφεληθούν από το μέσο αυτό επενδύσεων, το, την πρωτοβουλία Juncker και μέσα σε αυτά εξετάζουμε πάντα τα πράγματα υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε καλύτερα, καλύτερες εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση των αποβλήτων ώστε όταν μια, η τελική πρόταση της Κομισιόν καθορίσει το πώς θα θέλουμε να προχωρήσουμε, ήδη θα έχουν δημιουργηθεί κάποιες υποδομές και όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουμε με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Αυτή είναι η πρόθεση της Κομισιόν. <clears throat> Αυτά μπορώ να σας μεταφέρω αυτή τη χρονική στιγμή. Όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες για τις εναλλακτικέ προτάσεις μας, γιατί αυτές οι προτάσεις ακόμα είναι υπό επεξεργασία. Προσπάθησα όμως να σας δώσω μια κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται το έργο της Κομισιόν, <clears throat> προς τα που θα αναπτυχθούν όλες αυτές οι Αλλαγέ και οι προσπάθειες και σας υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν έχει κάνει μια πρόταση, ότι η τροποποιημένη πρόταση θα εμφανιστεί στα χέρια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου μέσα στο 2015. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για αυτήν την ε, παρουσίαση της κατάστασης. Πρέπει να πω προσωπικός και πριν αρχίσουμε να ακούμε τους συναδέλφους συντονιστές και τις ερωτήσεις τους. Μια μικρή παρατήρηση προς εσάς, κύριε Διευθυντά, από μένα. Είχα την εντύπωση από την παρέμβασή σας ότι βρισκόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Δηλαδή, βλέπω να υπάρχει μια αλλαγή στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προσθέσω ότι σε, όλες τις, σε όλα τα εγχειρίδια λογικής λέγεται ότι αν κάποιος λάβει μια απόφαση και την μεταβάλλει πρέπει και να αιτιολογήσει την αλλαγή. Ακόμα δεν έχω καταλάβει λοιπόν τους λόγους, τα αίτια. Θα θέλαμε αυτό να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα όλοι μας, διότι είναι σαφές ότι εάν Υπάρχει κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη την Επιτροπή ω προ την πρόταση και γι' αυτό θέλει να την τροποποιήσει. Να καταλάβουμε ακριβώ ποιο είναι αυτό το στοιχείο, ποια τα στοιχεία που δεν σα βρίσκουν σύμφωνους, που δεν αρέσουν πια στη νέα Επιτροπή. Αυτό πίσω από τα λόγια, καλύτερη νομοθεσία ή φιλοδοξότερο, δεν το καταλαβαίνουμε. Βεβαίως θα το ρωτήσουμε και στον ίδιο τον Επίτροπο και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα συναντηθούν μαζί μας εδώ στο επίπεδο αυτής της Επιτροπής. Όμως τα μέλη αυτής της Επιτροπής θέλουν να καταλάβουν τα αίτια. Διότι μόνο αν γνωρίζουμε τα αίτια μπορούμε να συμφωνήσουμε ή προφανώς να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Πάντως, ξεκινώ αμέσως δίνοντας το λόγο στους ε, συντονιστές ή τους εκπροσώπους τους ξεκινήσω από τον κύριο Φλόρεντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή νιώθω κάπως άβολα γιατί έχω ενώπιον μου ένα εξέχοντα υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επιτεθώ. Δεν με ικανοποιεί καθόλου κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε εδώ ένα υψηλό αξιωματούχο και όχι τον αρμόδιο επίτροπο. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα θέμα το οποίο ήταν τόσο αμφιλεγόμενο <clears throat> στην Επιτροπή μας και εδώ δεν ήρθε ο αρμόδιος επίτροπος ενώπιόν μας. Αν ήταν κάποιος ο οποίος δούλευε σε μια εμπορική επιχείρηση και δεν ήταν παρόν εδώ, θα τον απέλει εγώ. Θα πρέπει ο αρμόδιος επίτροπος να έρθει γιατί βρισκόμαστε σε αυτές τις δυσκολίες. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι καταπραϊντικά τα επιχειρήματα που μας έδωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αν πράγματι είναι τόσο φιλόδοξη η νέα Κομισιόν, δεν είναι τρόπος αυτός με τον οποίο αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο. Γιατί η προηγούμενη Κομισιόν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό επί τέσσερα χρόνια, έκανε 30 ή παραπάνω μελέτες που φαίνεται ότι ο αρμόδιος αντιπρόεδρος ούτε καν τις διάβασε. Και τώρα μέσα σε ένα χρόνο θα τροποποιηθούν όλα αυτά. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ θα ήθελα να πω ποια είναι η δική μου θέση εδώ. Εμείς δεν είμαστε κρατικοί υπάλληλοι. Είμαστε ευρωϊπάλληλοι οι οποίοι έχουμε εκλεγεί για να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Εγώ είμαι έτοιμος να εργαστώ με αυτό το φάκελο, αλλά όταν έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς η Κομισιόν βρήκε μια νομική βάση για να αποσύρει αυτή την πρόταση. Δεν είμαι νομομαθής, αλλά θα ήθελα να είναι εδώ ο Επίτροπός μας να μας εξηγήσει γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για να υπάρξει μια καλύτερη πρόταση. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε εμείς να θεσπίσουμε ε, στόχους ε, ε ανακύκλωση που να είναι ήδη μεταξύ Ρουμανίας και Αυστρίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το δεχτούμε. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κάποια διαφορά ακόμα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και Γερμανίας και Ιταλίας. Είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ίδια ε, ένωση και δεν μπορούμε εμείς να κρυπτόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πρέπει να έχουμε μια λύση η οποία να είναι ενιαία. Και πρέπει να ξεχάσουμε ότι με τις νέες ενέργειες που έχουν γίνει για την ε, εκλογή της Κομισιόν έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εκλέγει την Κομισιόν. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες είναι υποψήφιες, υπήρξαν υποψήφιες για την ε, Προεδρία της Κομισιόν, υπήρξε μια πίεση από την κοινή γνώμη. Και μετά έρχεται η Κομισιόν και λέει θα διαγράψουμε τις προτάσεις α, β, γ, δ κτλ. Πρέπει να έρθει εδώ όμως ο αρμόδιος αντιπρόεδρος και να μας εξηγήσει σε εμά και μέσω ημών στους εκλογείς μας γιατί παίρνονται τέτοιες αποφάσεις. Και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε τον ε, Καρλ Χάινς. Ο κύριος Δεμεσμάκερ. Ε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Είμαι σκιώδης εισηγητής. Με αυτή την ιδιότητα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε για αυτή τη συμβιλική κάπως παρουσίασή σας. Σε κάθε περίπτωση Καταντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε τα χαρτιά σας, όλα τα χαρτιά σας. Ε, αλλά παρόλα αυτά θα εκτιμούσαμε περισσότερες πληροφορίες. Θα ήθελα να απηχώντα την παρέμβαση του κυρίου Φλόρενς να προσθέσω και εγώ, ε, κύριε Φάλκινμπεκ, ότι ε, εγώ εξελίγνω στη Φλάντρα και εκεί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της ανακύκλωσης ε, και μάλιστα είμαστε πρωτοπόροι ε, σε θέματα που σχετίζονται με την ε, κυκλική οικονομία. Σίγουρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία για να σημειωθεί πρόοδος για κάποια από τα πιο βαρύνοντα ζητήματα. Ελπίζω ότι με τις τροπολογίες θα καταλάβετε πέραν κάθε αμφιβολίας πως ε, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως κάθε προσπάθεια που προωθεί την κυκλική οικονομία. Ας επανέλθω τώρα στην παρέμβαση του κυρίου Φλόρενς. Τα επιχειρήματα υπέρ αυτού του πακέτου μέτρων ε, είναι πιστικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα επιχειρήματα για την άρση αυτού του πακέτου μέτρων. Και Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ξεκάθαρη η πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων ή δεν θέλετε να βάλετε πολύ ψηλά τον πύχη διότι το σημείο εκκίνησης για κάποια κράτη-μέλη είναι χαμηλό. Είναι συγκεχημένο το μήνυμα που μας περνάτε. Επικρατεί σύγχυση σε σχέση με τα μέτρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης ε, με ποιο τρόπο ε, προτίθεστε να υλοποιήσετε εσείς αυτά τα μέτρα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις σας οι δικές μας. Είναι να προχωρήσουμε, να βελτιώσουμε τις προτάσεις που υπάρχουν. Φυσικά επιδέχονται βελτίωση και Είμαστε στο πλευρό σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία μας. Ε, κύριε Φάλκεμπερκ, ε, στις 4 Μαρτίου σας προσκαλούμε ήδη για μια ημέρα όπου θα γίνει επίδειξη στην Αμβέρσα και σε άλλες πόλεις ε, για τις ευέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία. Είναι καλό να δείξουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του πακέτου μέτρων ε, για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες επιδείξεις. Ε, είστε ευπρόσδεκτος κύριε Φάλκνερ και το ίδιο και ο Επίτροπος. Λοιπόν, θα συμπαραταχθώ με τον κύριο Φλόρεντς. Είναι εξαιρετικά λυπηρό που απουσιάζει ο Επίτροπος και δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το πακέτο μέτρων. Ευχαριστούμε η κυρία Κονέτσικα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονοματός ε, του συναδέλφου. Δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια ε, λόγω κάποιου κολλήματος ε, θα μιλήσω εγώ εξ ονόματος του συναδέλφου, εξάλλου ομονοούμε όλοι στην ομάδα μας. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό το πακέτο που μας προτείνετε, δεν το καταλαβαίνουμε στα πλαίσια της παρουσίασής σας. Ε, λέτε ότι θέλετε μέχρι το πέρας του έτους να καταθέσετε μία πιο φιλόδοξη πρόταση. εννοείται ακριβώς σε σχέση με το τωρινό πακέτο θα είναι λιγότερο φιλόδεξη η πρόταση. Η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σε όλους γνωστή. Αυτή η συμπεριφορά αποδεικνύει ότι τελικά θα χαμηλώσει ο πύχης. Θα είναι λιγότερο φιλόδοξο το νέο πακέτο που θα ενταχθεί στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι υποχρεωτικό ως εκ τούτου και πρέπει να σεβαστεί αυτή την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει βάσει του ε, εβδομού πακέτου πλαίσιο. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως υιοθετεί από τη φαίνεται μια διαφορετική προσέγγιση το Κοινοβούλιο, αλλά και το Συμβούλιο, αλλά ολόκληρη η κοινωνία των πολιτών υποστηρίζουν αυτό το πακέτο, διότι ενδιαφέρονται για το πώς διαχειριζόμαστε τα απόβλητα. Είναι ευρύτατη τη συνέντευξη στην οποία είχαμε καταλήξει και τώρα εσείς παραβλέπετε τα συμπεφωνημένα. Από πλευράς της GUNGL σας ε, δηλώνουμε με σαφήνεια ότι είναι δεν μπορούμε να δεχτούμε την απόσυρση αυτού του πακέτου για την παρουσίαση νέας πρότασης. Αυτό σημαίνει ότι όλη η δουλειά που έκανε ο κύριος Ποτόσνικ δεν θα ληφθεί τελικά η υπόψη. Έχουν γίνει συζητήσεις, διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες, με τους πολίτες, με τους ερευνητές και τώρα. Θα καταθέσετε μία νέα πρόταση ε, και δεν θα μπορέσουμε, σας το λέμε ήδη, δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με αυτή την πρόταση. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνει μια υποχώρηση. Αν δεν το κάνετε αυτό θα χάσετε κάθε αξιοπιστία ενώπιον του Κοινοβουλίου αλλά και της κοινωνίας των πολιτών διότι ξαναλέω όλοι συμφωνούν με αυτό το πακέτο. Προσοχή, είναι εξαιρετικά λεπτό το θέμα, μην υποτιμάτε τι συνέπειε των πράξεών σας. Ευχαριστούμε κύριε Γκεμπράντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη που έχω καθυστερήσει λιγάκι γιατί το τρένο μου καθυστέρησε. Νιώθω ακόμα σύγχυση σε σχέση με τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το πακέτο αυτό για τα απόβλητα και σε σχέση με την αντιμετώπιση της για την κυκλική οικονομία. Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε από την αρχή αυτής της συζήτησης όταν ήταν οι πρώτες φήμες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μπορεί να αποσυρθεί αυτό το νομοθέτημα, εμένα μου φάνηκε ότι υπήρχε έλλειψη επιχειρηματολογίας και έλλειψη πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξηγήσει γιατί ήταν γιατί πρόκειται να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει κάποιο ισχυρό, έγκυρο επιχείρημα που να εξηγεί γιατί πρέπει να αποσυρθεί το πακέτο για τα απόβλητα. Ο κύριος Τίμερμανς ήρθε στην ομάδα μας προσπαθώντας να το εξηγήσει, αλλά δεν είχε να μας προσφέρει κανένα επιχείρημα. Μιλούσε για την κυκλική οικονομία, που αυτό το πακέτο αντιμετώπιζε μονάχα το ίμιση του κύκλου και μετά μίλησε για την επαναχρησιμοποίηση που δεν περιλαμβανόταν μέσα σε αυτό το νομοθέτημα και την ε, περιεκτικότητα σε άνθρακα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί χωριστά. Κανένας που ξέρει το θέμα αυτό δεν κατάλαβε μία για αυτά τα οποία είπε. Ούτε και οι υπόλοιποι φυσικά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν καταλαβαίνω την βάση για αυτή την απόσυρση, την επιχειρηματολογία. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολιτικούς λόγους θέλει να δείξει στον κόσμο την έτοιμη να υποσκάψει το ε, κοινοτικό κεκτημένο, τουλάχιστον να το κρατήσει εκεί που είναι και να μην το διευρύνει περισσότερο και να αρχίσει να ακυρώνει διάφορα νομοθετικά στοιχεία. Αυτό, το, αυτό δεν το είπε ο κύριος Στίμερμαν στην πολιτική μας ομάδα, αλλά αυτό ακούω τώρα να αναφέρεται από διάφορες φήμες, ότι δεν είχε αρκετά οικονομική εστίαση το πακέτο αυτό. Αλλά μα δείτε την πρόταση την ίδια. Ξεκινάει αναφερόμενο στην οικονομία. Μιλάει για εξοικονομίες 600 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο άλλο τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να εξοικονομήσουμε τόσα πολλά χρήματα για τι βιομηχανίε μα. Η έλλειψη λοιπόν οικονομική επιχειρηματολογία δεν ήταν το πρόβλημα. Αυτό θα έπρεπε να ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της νέας πρότασης για να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Τα έχω χάσει λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Το μόνο πράγμα το οποίο θα δούμε τώρα είναι ότι μάλλον θα δαπανίσουμε πολύ χρόνο, ίσως ένα χρόνο, μπορεί να είναι και δύο χρόνια, τον Ιούλιο παρουσιάστηκε αυτή η πρόταση στο Κοινοβούλιο. Εμεί δεν μπορούμε να περιμένουμε να υπάρξει μια νέα πρόταση μέχρι το τέλο του τρέχοντο έτου. Αυτό λοιπόν <clears throat> θα σημάνει μια καθυστέρηση ουσιαστικά δύο ετών. Και δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα, δεν είναι μονάχα η καθυστέρηση. Αυτό το οποίο ακούω τώρα είναι ότι όταν θα αντιμετωπίσει η δια υπηρεσιακή ομάδα της Κομισιόν αυτή την πρόταση, θα καταλάβουν ότι είναι πολύ δύσκολο να προτείνουν οτιδήποτε καινούριο το οποίο μπορεί να, να διαφοροποιηθεί από την τωρινή πρόταση. Η Κομισιόν δηλαδή θα προσπαθήσει απεγνωσμένα να βρει νέα στοιχεία να βάλει στη νέα πρόταση και αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ποιότητα της πρότασης αυτής. Για μια ακόμα φορά λοιπόν θέλω να κάνω μια έκκληση προς την Κομισιόν να ξανασκεφτεί για τη στρατηγική της. Δεν θα πούμε ότι είναι μεγάλη ήττα της Κομισιόν όταν ξανακαταθέσουμε μια πρόταση σε δύο μήνες με ουσιαστικά επιφανειακές αλλαγές. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και η οικονομία πρέπει να κερδίσουν και αυτό είναι για το οποίο πρέπει εμείς να αγωνιστούμε. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Σλέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Φάλκενμπεργκ. Λυπούμε πολύ που βλέπω ότι το πακέτο αυτό αποσύρεται από την νομοθετική διαδικασία. Βρίσκω ότι είναι μεγάλη καθυστέρηση αυτή σε σχέση με όσα έχουν γίνει τα περασμένα ε, χρόνια με τόσες προσπάθειες από το Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τον ε, Επίτροπο Ποτότσνικ. Ο σκοπός ήταν να προσαρμοστεί στις ανάγκες μας όλο αυτό το πακέτο με τόσες προτάσεις. Να ε, επισημάνω ότι τη φτάση της αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ευθύ εξ αρχής ότι το περιβάλλον είναι ένα μαύρο πρόβατο στο σύνολο της θητείας της Επιτροπής για αυτό το διάστημα, διότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι κάτι που σχετίζεται μόνο με την οικονομία, αλλά πρωτίστως με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί είναι ότι ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ή μάλλον σκοπεύει να υποβάλει φιλοδοξότερες προτάσεις. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν σχόλια, παρατηρήσεις και αντιρρήσεις ως προς το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι υπερβολικά φιλόδοξο ως προς την σταδιακή ε, εξάλληψη των χωματερών. Η πρόταση λοιπόν, ε, υπόσχεση αυτή ότι είναι πιο φιλο... θα είναι πιο φιλόδοξες οι προτάσεις της Επιτροπής που θα έρθουν για να συνδυαστεί με την κυκλική οικονομία, αυτό αντιφάσκει μόσο από από ο κ. Γιούνκερ στην προκλογική του εκστρατεία. Ε, εντόπισε το, πακέτο αυτό κάτι αρνητικό και ως ένα άχθος, ε, ένα πρόβλημα για το όλο σύστημα. Τέλος, να πω ότι να το πω και να το πω αρκετά έντονα ότι το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσύρει αυτό το πακέτο δεν μπορεί να είναι θετικό ως μήνυμα. Είναι πολλές οι χώρες που φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν ούτως ή άλλως να καλύψουν το στόχο της εξέλιξης των χωματερών. Αυτή σας η κίνηση τους δίνει την εντύπωση ότι μπορούν να παραμείνουν στις ίδιες διαδικασίες. Ευχαριστώ η συνάδελφος Εύη. Ευχαριστώ να συμφωνήσω με τα σχόλια των συναδέλφων. Οπωσδήποτε η απόφαση απόσυρσης του πακέτου δεν είναι καθόλου θετικό μήνυμα για την έναρξη θητείας και ανάληψης καθηκόντων της Νέας Επιτροπής. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τους συναδέλφους και να πω ότι ο Επίτροπος Βέλα θα έπρεπε να είναι εδώ για να μας δώσει μια απάντηση. Και όχι μόνο επειδή το κόστος που ε, έχουν ε, φέρει τόσες μελέτες, η μελέτη αντικτύπου, ε, όλες οι έρευνες, με δημόσια έγιναν όλες αυτές. Θα έπρεπε να το έχουμε και αυτό κατά νου. Επίσης να τονίσω ότι σε αυτή τη φάση, στη νέα πρόταση, δεν μπορεί να δοθεί περισσότερος χώρος για καλύτερες εξελίξεις σε κάποια σημεία. Όπως η συγκεκριμένη κοστολόγηση των αποβλήτων. Αυτή η επιλογή που θα δώσει συνέχεια στην αρχή του «Ρηπαίνων πληρώνει» θα συμπεριλάβει και τα βιολογικά απόβλητα πλέον. Κάτι εξίσου σημαντικό για να ασχοληθούμε με την διαχείριση των αστικών αποβλήτων με το σωστό τρόπο. Και Ολοκληρώνοντας μια τελευταία παρατήρηση για το μοντέλο, το μοντέλο των αποτεφρωτών, των αποβλήτων, της καύσης των αποβλήτων, των σκουπιδοφάγων στην ουσία, που δεν επιτρέπουν ουσιαστικά τη μείωση, τον περιορισμό των αποβλήτων μελλοντικά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θεωρήσουμε σώρευση αποβλήτων που νομίζω ότι στην κοινωνία μας είμαστε αναγκασμένοι να την ε, υποστούμε και θα τη συνεχιστεί. Η καύση λοιπόν χρησιμοποιείται κυρίως με αποτεφρωτές. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση. Πρέπει να σκεφτούμε και άλλες επιλογές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τους σκιώδεις εισηγητές και τις ερωτήσεις τους. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο και στους συναδέλφους για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, παρακαλώντας να είστε σύντομοι. Ματίας. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ο κύριος Γιούνκερ είχε πει ότι θέλει μία πολιτική επιτροπή και πολλοί το έχουν επικροτήσει αυτό και σήμερα τώρα του επιτίθενται πολλοί γιατί δεν έχει πραγματικά κάνει κάτι διαφορετικό, παρά μόνο μια πολιτική απόφαση. Ορισμένοι λένε ότι αυτό γίνεται από την πίεση των ε, λόμπι. Και καλώς ήλθαν και τα λόμπι εδώ στην αίθουσα που είναι παρόντα εξάλλου. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας αφήνει εμβρόντιτους ότι αντιμετωπίστε μια πρόταση με τον τρόπο αυτό. Τι γίνεται με την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει. Το να αποσυρθεί αυτό το πακέτο γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν ευνοεί τις επενδύσεις και την βιωσιμότητα των επενδύσεων. Και εγώ ως ε, προεχόμενος από τη Φριζία ε, ενοχλήθηκα από αυτά που ελέγχθηκαν στα Ολλανδικά διότι τα κατανοώ από τον κύριο Τίμερμανς και εγώ ενοχλούμαι από αυτά που έκανε ο κύριος ε, Τίμερμανς από την πλευρά της Κομισιόν. Αυτό δεν έχει ενισχύσει καθόλου την ε, εμπιστοσύνη προς την Κομισιόν και αυτό είναι ένα ουσιαστικό θέμα σε ό,τι αφορά τους επενδυτές να υπάρχει μια εμπιστοσύνη αυτού του είδους. Αυτό είναι ένα αράπισμα λοιπόν το οποίο μας δόθηκε από την Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Εμείς περιμένουμε να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία θα σκεφτεί και το θέμα της βιωσιμότητας. Η καμπύλη μάθησης νομίζω ότι πρέπει τώρα να έχει φτάσει στο υψηλό της επίπεδο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε η Κομισιόν τώρα θα καταλάβει πού κάνει λάθος. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό σε μια χρονική στιγμή που έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα από το να κοιτάμε αν πρέπει να αποσυρθεί ή όχι μια πρόταση. Μια πρόταση δεν είναι ποτέ τέλεια αλλά γι' αυτό υπάρχει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να βελτιωθούν οι προτάσεις. Τι νόημα έχει αυτό να προσπαθεί η Κομισιόν να τα κάνει όλα τέλεια όταν υπάρχει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που θα πρέπει να επεξεργαστούν αυτό το πακέτο. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να ευσταθεί το επιχείρημα αυτό ότι δεν είναι αρκετά καλή αυτή η πρόταση και να κάνουμε μια καλύτερη πρόταση. Δεν υπάρχει χειρότερο επιχείρημα με τον τρόπο αυτό φανταστείτε τι θα κάνει οι Υπουργοί Εξωτερικών αν είχαν να αντιμετωπίσουν θέματα όπω τη Παλαιστίνη ή τη Ουκρανία και να λέγανε Α, αυτή η πρότασή μα δεν είναι καλή, θα την αποσύρουμε, θα ξαρχίσουμε από την αρχή. Λοιπόν, δεν έχουμε με τον τρόπο αυτό καμία δυνατότητα να προχωρήσουμε. Και αυτό το οποίο έχει κάνει η Κομισιόν ουσιαστικά έχει υπονομεύσει τη θέση τη. Στο Ματία η κυρία Άουκεν. Μα σα παρακαλώ, να είστε σύντομοι γιατί αλλιώς θα έχουμε δυσκολίες για την ακρόαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πραγματικά ποιον προσπαθείτε να κοροϊδέψετε κύριε Φάλκινμπεργκ. Ε, ξέρετε, πολύ καλά πόσο αγωνίστηκε για χρόνια ολόκληρο ο Επίτροπος Ποτόσνικ ε, για αυτό. Και εδώ μας λέτε, έρχεστε εσείς σήμερα και μας λέτε θέλω, θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος ακόμη έχετε υποβαθμίσει τη σημασία του περιβάλλοντος ε, στην ε, Επιτροπή. Τίποτα δεν κάνετε για να κάνετε τα λόγια πράξη. Α, το eco-design θα μου πείτε. Ξέρετε ότι ο Γιούνκερ έκανε καμπάνια κατά την προκλογική του εκστρατεία κατά της οδηγίας για το οικολογικό ε, design. Συγγνώμη, ε, να μας τα λέτε λίγο πιο ξεκάθαρα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, διότι ε, δεν ωφελεί να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι. Κανείς δεν θα αποκομίσει κάποιο όφελος έρχεστε συνήθως και μας λέτε ότι ε, είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι και τώρα σε τι παιχνίδι παίζετε. Έρχεστε και μας λέτε ότι εσείς θέλετε να είστε ακόμη πιο φιλόδοξος ε, και τι έχετε, θέλετε να μας πείσετε ότι έχει προσιλητιστεί στα περιβαλλοντικά ζητήματα ξαφνικά ο κύριος Γιονκέρ. Ε, ξέρετε ότι ε, λέμε κάτι στα δανέζικα. Το νόημα είναι ότι θα πρέπει να πείτε στον πρόεδρό σας ότι πρέπει τουλάχιστον να σώσει την εικόνα του γιατί έτσι μπορεί να σώσει και τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ποκ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι γνωστό ότι είμαι Συνήθως ε, ε, στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Φάλκενμπερκ ξέρει ότι υποστηρίζω συνήθως την Επιτροπή. Κύριε Φάλκενμπερκ, όμως ε, σήμερα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή γιατί είναι γνωστά αυτά τα ζητήματα που συζητούμε και αν η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλει να υποκύψει στην πίεση αυτών που δεν θέλουν να επενδύσουν, δεν θέλουν να κάνουν τις καινοτομίες ε, και θέλετε να γνωρίζετε τις κίτρινες κάρτες ε, που κραδένουν πολλά εθνικά κοινοβούλια ήδη, δεν θα πρέπει να ξαφνιαστείτε με αυτά που θα συμβούν στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Εμείς ε, θέλουμε να διατηρηθεί το πακέτο για τα απόβλητα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πολύ αμφιβάλλω εάν ε, ε, είναι σε θέση καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Η κυρία Όκεν ε, πολύ καλά το είπε, ας μην ε, βαφκαλιζόμαστε, ας πούμε ξεκάθαρα περί ως πρόκειται και ε, ας μην υποκύψουμε στην πίεση αυτών ε, που στον τομέα της βιομηχανίας ε, που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Ε, θα αρχίσει πόλεμος ανάμεσα στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου λόγω αυτού του πακέτου. Αν συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε. κυρία... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οδηγία η οποία προτείνεται αφορά ένα θέμα στο οποίο εγώ αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχει να κάνει με την ικανότητά μας να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ε, πόρους που αποκτούμε από τη, από τη φύση και να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά δεν θα εκπλήξω κανένα όταν λέω ότι η ανακύκλωση είναι ένα τεχνικό και τεχνολογικό θέμα. Γι' αυτό πολλά κράτη και δήμοι και τοπικές κοινότητες αναθέτουν αυτό το έργο σε ειδικευμένε επιχειρήσεις. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αυτό συναρμόζεται με ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και πρότυπα για τις επιχειρήσεις και, τους, και οι δήμοι. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις σε επίπεδο και προϋπολογισμού. Θα πρέπει να δημιουργήσουν να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις και αυτό σημαίνει και μια βαθιά εκβάθρων αναδιοργάνωση της οικονομίας μας και τη της βιομηχανίας μας. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να προχωρήσει σε μια συνολική αξιολόγηση, έγιναν τέτοιες αξιολόγηση, αλλά δεν είναι επαρκή, να υπάρξει πραγματικά μια αξιολόγηση αντικτύπου για τις συνέπειες που θα προκύψουν για μια κυκλική οικονομία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αποδοτική με μια τέτοια οικονομία. Υπάρχουν μεγάλες ανισομέρειες μεταξύ των κρατών μελών που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Τα κράτη-μέλη ίσως είναι πολύ καλύτερα να επιφέρουν αυτή την αναδιοργάνωση που απαιτεί η κυκλική οικονομία καλύτερα από την Κομισιόν. Ο κύριος Πέτρελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα απόβλητα είναι ένα από τα κομβικά κοινά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να το πράξουμε αυτό όμως, πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα. Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να γίνουν απόβλητα και από τις πολιτικές συζητήσεις. Θα ήθελα να υπάρξει μια δεσμευτική απόφαση η οποία να καθορίζει τους σαφείς στόχους και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Δεν πρέπει να έχουμε ασυνέχειες σε νεολογικό επίπεδο. Δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να υποστηρίσουμε την κυκλική οικονομία και σε μια μεταγενέστερη συνεδρία να υποστηρίσουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Η φιλοσοφία που είχε η προηγούμενη Κομισιόν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, τη διαχείριση των αποβλήτων, πιστεύω ότι ήταν μια σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εδώ έχουμε ενώπιον μας ένα πολύπλοκο θέμα. Μια καθαρά τομεακή αντιμετώπιση δεν θα μας πάει πολύ μακριά. Χρειαζόμαστε μια συνολική αντιμετώπιση η οποία θα ενσωματώσει όλες τις πτυχές αυτές. Κάτι ακόμα. η πολιτική μας για τα απόβλητα όλη, αυτή η πολιτική έχει να κάνει με το ένα στόχο που συμμεζόμαστε με την ευρωπαϊκή οικονομία μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Θα ήθελα να έχω περισσότερες απαντήσεις από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Φλάναγκαν τώρα. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλούς διερμηνείς στην, σε όλες τις ε, <laughs> επιτροπές, αλλά φαίνεται ότι μας λείπει μία γλώσσα ε, τη, τα τεχνοκρατικά, τα τεχνοκρατικά για να τα μεταφράσει ναι. Ε, πρόκειται για κορακίστικα που δεν καταλαβαίνουμε. Ε, ξέρετε, ε, ό,τι κορακίστικα και να μιλάτε, ε, εγώ, ξέρετε πώς το μεταφράζω αυτό που λέτε στο μυαλό μου, δεν σε εμπιστεύομαι, δεν εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεκάρα τσακιστή δεν δίνεται για το περιβάλλον. Και γι' αυτό είναι καταστροφή αυτή η νέα Επιτροπή του Γιούνκερ και πρέπει να αποπέμφθει. Ε, σας ευχαριστούμε. Ε, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις απαντήσεις. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή όλες ε, τις διαφορετικές απόψεις και σε μεγάλο βαθμό νομίζω πως επαναλαμβάνουν θέσεις που έχουμε ακούσει και σε προηγούμενες συζητήσεις, συγκεκριμένα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Ε, ξέρετε, για πολλούς λόγους δηλώνει ικανοποιημένος <laughs> για την ε, ε, υποστήριξη για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι προηγουμένου. Τέτοιον ενθουσιασμό δεν τον έχω ξαναζήσει. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, ε, αλλά μία διαλέξαμε να την αποσύρουμε για να τη βελτιώσουμε, έτσι. Και ξαφνικά ε, δεν ε, έχει υπάρξει τόσο μεγάλος ενθουσιασμός για αυτή την πρόταση που θέλουμε να αποσύρουμε. Το ίδιο σημαίνει και στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο όταν δεν ήξεραν ακόμη ότι ενδεχομένως και να την αποσύρουμε, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για το περιβάλλον είχαμε ε, ένα πολύ μεγάλο κατάλογο ερωτήσεων και επικρίσεων ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο, ότι είναι υπερβολικά περίπλοκο μας έλεγαν, ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό και ε, ήταν ατελείωτος ο κατάλογος με τα κατηγορώ. Παρόμοιες αντιδράσεις λοιπόν έχουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε επαφές που έχω με ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και άλλων ενώσεων. Η τωρινή πρόταση φυσικά γίνεται πλέον πολύ καλύτερα αντιληπτή σε σχέση με κάτι το άγνωστο και ε, την χάνει μεγάλης υποστήριξης, ευρείας υποστήριξης. ξέρετε, είναι πλάκιν ανάμεσα στη σύνταξη ε, της υφιστάμενης πρότασης ε, και δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι τέλεια και ότι δεν ε, επιδέχεται βελτιώσεις. Κάποια από τα σημεία ήδη τα σχολιάσατε. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτι που δημιουργεί εμπιστοσύνη για τους επενδυτές και να βασίζεται αυτή η πρόταση σε μια βασική περιβαλλοντική ανησυχία. Στην, αναφέρθηκα στην ανάλυση της ε, αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, ε, ε, μια έννοια στην οποία εδράζεται η πρόταση, αλλά χρειαζόμαστε να κατοχυρώσουμε και την οικονομική βιωσιμότητα αυτής της πρότασης με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Άκουσα πολλά σχόλια για το ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τους ε, χίτα σε, αυτό, σε τόσο μεγάλο βαθμό ε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως input για την επόμενη γενιά προϊόντων, ότι πρέπει να αποφεύγουμε την ε, παραγωγή αποβλήτων, να επιδιορθώνουμε τα προϊόντα αντί να τα απορρίπνοντα στους χίτα όπως συχνά γίνεται τώρα και αυτή την επιχειρηματολογία την έχω ακούσει ήδη σε επίπεδο κρατών μελών και είναι χειρότερη. Την ακούω και εδώ. Παραμένει όμως το δεδομένο ότι ένας μεγάλος αριθμός κρατών μελών διαθέτουν 90% των δημοτικών αποβλήτων τους σε χήτα. Ναι, η Φλάνδρα Πολύ ωραία. Έδειξε ταχύτατα ότι μπορούμε να αλλάξουμε πορεία, ότι υπάρχουν τρόποι ε, να, για να μετατρέψουμε μια γραμμική οικονομία σε κυκλική, ε, χρησιμοποιώντας ε, διαφορετικές ε, ροές αποβλήτων. έχω ήδη επισκεφθεί πολλές επιχειρήσεις στη Φλάνδρα και ξέρω ότι ε, γίνεται πάρα πολύ έρευνα, κοινοτομία, δράσεις, πρωτοβουλίες ε, για την ανακύκλωση του PVC και άλλων ε, μορφών πλαστικού υπάρχουν πολύ καλά, πολύ ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης για τέτοιου είδους ροές αποβλήτων. Παρόλα αυτά, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν Ισχύει αυτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να αναρωτηθούμε γιατί κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατορθώσει τελικά να μειώσουν τον αριθμό των, αποβλήτων, ε, των δημοτικών αποβλήτων στους ε, ΧΙΤΑ και να περιοριστεί ε, στο 1-2% και άλλοι πάλι είναι στην άλλη άκρη της ψαλίδας και έχουν φτάσει μέχρι και το 95%. Έγινε αποτίμηση των προτάσεων και το υλικό που έχουμε επεξεργαστεί και στο οποίο έχουμε καταλήξει δεν χάνεται. Δηλαδή η ανάλυση που έχουμε κάνει και το προϊόν της ε, ε, ε, στο οποίο βασιζόταν η πρότασή μας παραμένει ακέραιο. Όμως χρειαζόμαστε καλύτερη κατανόηση. Γι' αυτό εισηγούμαστε μια νέα πρόταση. Υπάρχουν νομοθετικές απαιτήσεις ε, για κάποια κράτη-μέλη το 2015 για την θέσπιση συστημάτων ε, ε, χωριστής συλλογής για να υπάρχουν ξεχωριστές ροές αποβλήτων για το πλαστικό, για το χαρτί, για το μέταλλο, για το γυαλί. Και για τα βιοαπόβλητα είναι ξεκάθαρη η γραμμή μας ότι δεν πρέπει να διατίθενται ανεπεξέργαστα στους χήτα. Παρόλα αυτά ε, εξακολουθούν να συμβαίνουν αυτά και αρχίσαμε μια αποτίμηση όπως σας έλεγα για να κατανοήσουμε καλύτερα ποια συστήματα ξεχωριστής ε, ε, συλλογής έχουν ήδη ε, θέσει σε λειτουργία τα κράτη-μέλη γιατί υπάρχει το 2015 η υποχρέωση συμμόρφωσης ε, και θέλουμε να ξέρουμε το 2015 ε, θα αρχίσει η διαφορετική συλλογή ούτω ώστε μέχρι το 2025 να μπορέσουν αυτές οι χωριστές ροές αποβλήτων να απορρίπτονται στους ΧΙΤΑ, όπως προβλέπετε για την τελική τους ε, διάθεση. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος ε, για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς ε, δε είπε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταθέσει μια πληρέστερη, πιο φιλόδοξη πρόταση. Μπορείτε όμως να την κρίνετε μόλις κατατεθεί. Δεν μπορείτε να κρίνετε κάτι που δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το στάδιο είναι ότι εργαζόμαστε με επικοδομητικό πνεύμα ούτω ώστε με αυτήν την πολιτική να συμβάλλουμε στην τόνωση της οικονομίας, στη δημιουργία των θέσεων εργασίας. Υπάρχει ε, ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό και ε, ταχύτατα μπορούμε να το απελευθερώσουμε με τέτοιου είδους ε, δράσεις. Δεν σχολίασα το περιεχόμενο και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω της οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε όμως ότι για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε χωρίς τα νομοθετήματα, έχουμε στόχους που έχουν ως χρονικό ορίζοντα το 2020. Πολλά κράτη-μέλη σε αυτό το σημείο δεν θα φαίνεται ότι θα είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους στόχους τους ε, το 2020 και με τη νέα πρόταση θέτουμε πιο φιλόδοξους στόχους ε, παρατείνοντας την προθεσμία το 2030. Αύριο το πρωί νυχθημερών δεν πρόκειται να ε, συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Όμως έχουμε το περιθώριο να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων και έχοντας ακούσει τις αντιδράσεις εδώ στο Κοινοβούλιο και τις αντιδράσεις των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει τη δέσμευση πριν ε, το τέλος του 2015 να καταθέσει μια πρόταση. Τώρα σε ποιους τομείς και πού θα είμαστε πιο φιλόδοξοι νομίζω ότι ε, σας έδωσα κάποια στοιχεία πού θα υπάρξουν νέες προτάσεις δηλαδή για τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων με τρόπο ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα στη συνέχεια οι προσπάθειες ανακύκλωσης. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ε, μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ όμως να σας πω ότι αναλύουμε τις πολύ διαφορετικές καταστάσεις που ε, υπάρχουν σήμερα στα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία ουσιαστικά θα μπορέσει να υλοποιηθεί από τα 28 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Δευθυντά. Καταρχάς ευχαριστούμε που δεχτήκατε να έρθετε στην Επιτροπή μας παρόλο που καλά γνωρίζατε τι είχε προηγηθεί στις συζητήσεις. Δηλαδή, ότι ουσιαστικά είχαμε εξελιχθεί σε μια αρένα ταυρομαχίας ε, εδώ και ότι εσείς δεν θα ήσασταν σίγουρα ο ταυρομάχος. Ο ταυρομάχος θα έπρεπε να είναι ο επίτροπος που θα περιμέναμε σήμερα εδώ για να μας δώσει λεπτομερείς εξηγήσει για τα αίτια της επιλογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο ε, της ημερής διάταξης που είναι η ακρόαση ακρόαση η οποία θα ε, οργανωθεί όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Να δώσω το λόγο στην, ε, στον εισηγητή και θα καλέσω όσους θέλουν να φύγουν από την αίθουσα να το κάνουν ησύχως για να μπορέσει ε, να ξεκινήσει γρήγορα η ακρόαση. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Η εισηγήτρια, κυρία Μποναθέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουμε σημαντικούς προσκεκλημένους, θα είμαι πολύ σύντομη. Στην παρουσίαση αυτής της ακρόασης. Γιατί οργανώσαμε την ακρόαση παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως τώρα. Είναι ένα θέμα συνέπειας και αξιοπιστίας. δεν ήμασταν εμεί ασυνεπεί στι υποχρεώσει μα, λιγάκι φάνηκε έτσι η Επιτροπή. Εμεί θα προχωρήσουμε με τι επιτάπητο προτάσει, ελπίζοντα να δούμε και την ουσία του θέματο. Οργανώσαμε λοιπόν αυτήν την ακρόαση σε δύο τμήματα. Πρώτα απ' όλα, για να δούμε ένα γενικό, ε, μια γενική εικόνα για την κυκλική οικονομία και μετά τα κρίσιμα σημεία της πρότασης. Γιατί το πρώτο τμήμα για την κυκλική οικονομία. Γιατί είναι σαφές ότι οδηγεί για τα απόβλητα είναι ένα απόσπασμα στο τμήμα της πρότασης για την κυκλική οικονομία. Όπως προέκυψε και από την συζήτηση που μόλις έγινε, φαίνεται ότι η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία έχει να κάνει και με την ε, ορθολογιστική χρήση των πόρων με υψηλότερους στόχους για την ε, ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τα απόβλητα που ίσως να μην ε, θεωρούνται πλέον ως τέτοια, αλλά ως αξία. Ως κάτι που μπορεί να αποφέρει κέρδος. Αλλάζει λοιπόν το μοντέλο που ίσχυε σήμερα. Σε πρώτη φάση λοιπόν αποφασίσαμε να συζητήσουμε από κοινού με τους βασικούς ενδιαφερομένους. Τους τελευταίους μήνες Συνάντησα πολλούς από τους ενδιαφερομένους του τομέα και κατάλαβα ποιες είναι οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες της πρότασης όπως παρουσιάζεται και πολύ γρήγορα επί της ουσίας η μέθοδος υπολογισμού είναι και μια από τις προστιθέμενες αξίες, ο γενναία μέθοδος υπολογισμού, αλλά συμπεριλαμβάνει και δυσκολίες. Πρέπει να καταλάβουμε τι θα υπολογίζουμε Ποιο είναι το κομμάτι της ανακύκλωσης, ο ορισμός των δημοτικών αποβλήτων που θα πρέπει να τον ξαναδούμε, το θέμα των ευθυνών των παραγωγών. Πιστεύω όμως ότι πέραν των συναντήσεων και συνομιλίων που είχα εγώ, αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να έχουμε και την άποψη των προσκεκλημένων μας. Περιορίζομαι λοιπόν στο καλωσόρισμα προς όλους και σας ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ. πολύ. Και τώρα ξεκινούμε με τις ε, παρουσιάσεις. Παρακαλώ να παραμείνετε στα 6 λεπτά ή δυνατόν από τον ε, Τζος Μπλέριοτ, ο οποίος είναι από το Ίδρυμα Έλεν Μακάρθου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. για το Ίδρυμά μου. Δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός. Είμαστε ένας φορέας ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια με το στόχο να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία τονίζοντας τις οικονομικές ε, ευκαιρίες οι οποίες θα δημιουργηθούν. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και με εκπαιδευτικά ιδρύματα για να μπορέσουμε να, ξε, να τονίσουμε την ανάγκη να περάσουμε από μια γραμμική οικονομία η οποία βασίζεται στην κατανάλωση των φυσικών πόρων σε μια κυκλική οικονομία η οποία εξασφαλίζει τη δημιουργία αξίας των φυσικών πόρων. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Υπάρχει φυσικά ένα σύνολο από παράγοντες που έχουν συνενωθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει η ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Η χρηματοπιστωτική και επενδυτική κοινότητα θέλει να βρει πιο σταθερές και πιο ανθεκτικές ευκαιρίες επενδύσεων. Ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη να βρούμε νέες ε, διεξόδους για την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης έχουμε και μια νέα μορφή καταναλωτή ο οποίος έχει αναδυθεί, ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο έχει πρόσβαση στους πόρους και τα προϊόντα και όχι να είναι ιδιοκτήτης τους, τον νοιάζει πιο πολύ να έχει τις υπηρεσίες από τα προϊόντα αυτό και αυτό δίνει πολλές δυνατότητες σε ό,τι αφορά την αμοιβεοποίηση των πόρων και των υπηρεσιών σε μια οικονομία και τέλος, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, υπάρχει και η ενηλικίωση κατά κάποιο τρόπο της τεχνολογίας πληροφοριών που μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τα υλικά και τους πόρους, να ξέρει από τι παράγεται το κάθε προϊόν και να ξέρει και πόσο, είναι, πόσο διαρκεί η χρήσιμη ζωή τους. Αν λοιπόν τη δούμε σαν γράφημα αυτή την κυκλική οικονομία, Ίσως δεν είναι ευανάγνωστο αυτό το γράφημα. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε εδώ μια συστημική αλλαγή. Έχουμε πολλούς οι οποίοι εμπλέκονται και πολλούς τομείς οι οποίοι εμπλέκονται. Αλλά έχουμε εδώ μια διάκριση μεταξύ βιολογικών υλικών από την μια μεριά και τεχνημάτων, τεχνικών υλικών. Και από την οικονομική μας ανάλυση είναι φανερό ότι η μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες για αξιοκονόμηση ενέργειας βρίσκονται περίπου <clears throat> στο κέντρο του γραφήματος σε ό,τι αφορά την αναχρησιμοποίηση στην ε, διαδικασία παραγωγής και την ε, επαναξιοποίηση. Όλες αυτές οι τεχνικές που επιτρέπουν επαναχρησιμοποίηση. Για παράδειγμα, αν πάρουμε το μπλοκ της του κινητήρα σε ένα αυτοκίνητο, ένα που έχει δημιουργηθεί από νέα υλικά και ένα το οποίο έχει ξεκινήσει από μία ανακύκλωση, το δεύτερο μας δίνει τη δυνατότητα μιας ε, εξοικονόμησης ενέργειας κατά 75% και αυτό φυσικά και θετικές συνέπειες <clears throat> για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως πρέπει να υπάρχουν και ορισμένες επιλογές σχεδίασης, να μπορούν να αποχωριστούν τα συστατικά στοιχεία του κινητήρα εύκολα, να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίηση των υλικών, να μην υπάρχει ρήπανση η οποία προκαλείται από αυτήν την ε, διαδικασία. Αν θέλουν ε, λοιπόν οι κατασκευαστές να χρησιμοποιήσουν τα υλικά τους αυτά ώστε να τα κρατήσουν ως βασικά υλικά και δεν χρειάζεται να έχουμε νέα ε, χρήση φυσικών πόρων, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το, <clears throat> ορισμένα μοντέλα επιχειρηματικά όπως είναι την, ε, για την πληρωμή, για τη χρησιμοποίηση ή το leasing. Το 2012 εκθέσαμε, παρουσιάσαμε μια έκθεση <clears throat> και είχαμε και την υποστήριξη της Κομισιόν για το θέμα αυτό ζήτησε η Κομισιόν από το Ίδρυμά μας να είναι ένας από τους εμπειρογνώμονες σε σχέση με την πλατφόρμα για την ε, αποτελεσματικότητα των πόρων. Είχαμε εμπλακεί λοιπόν στις συζητήσεις αυτές σε σχέση με το πακέτο κυκλικής οικονομίας και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μας. Αυτή η πρώτη έκθεση λοιπόν κατέδειξε και νομίζω ότι είχε αναφερθεί αυτός ο αριθμό ότι υπάρχει μια δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή ε, μεταπηδική οικονομία για προϊόντα όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα οικιακά ηλεκτρονικά, τα πλυντήρια κτλ. μπορούν να προκύψουν κάτι μεταξύ 400 και 630 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο σε επίπεδο εξοικονόμησης και αυτό βλέποντας μονάχα τις δυνατότητε να αλλάξουμε τις ε, προδιαγραφές σχεδίασης. Δεν πρόκειται για κάτι το επαναστατικό. Αυτό για να σας τονίσω ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία, μπορούμε να την αδράξουμε και με το να διευρύσουμε τις κατάλληλες συστημικές ε, ευκαιρίες στο συστημικό πλαίσιο μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα και κάποιες επιχειρήσεις ήδη αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτές τις ευκαιρίες. Είναι λοιπόν θέμα του να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις, τα σωστά μηνύματα προς τους επενδυτές για να ευνοήσουμε αυτά τα κυκλικά συστήματα παραγωγής και όχι το γραμμικό σύστημα το οποίο έχει τα γνωστά μειονακτήματα και ιδίως στη δημιουργία αποβλήτων. Έρχομαι λοιπόν στο τέλος των έξι λεπτών. Απλώς θέλω να, να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα. Η δεύτερη έκθεση την οποία εμείς έχουμε δημοσιεύσει αφορά ορισμένα πιο βιολογικού χαρακτήρα αγαθά. Και εδώ μπορούν να γίνουν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά το κλείσιμο του βρόχου για τις, ε, τα διατροφικά προϊόντα και έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες που τα χρησιμοποιηθούμε και να αντιμετωπίσουμε επίσης και το θέμα της ε, απώλειας τρεπτικών ουσιών στο έδαφος. Υπάρχουν πάρα πολλά για να κλείσουμε το βρόχο και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα σωστά αγροτικά προϊόντα τα οποία επανέρχονται μέσα στο σύστημα. Κατά τη δική μας άποψη λοιπόν είναι ε, ένα θεματολόγιο το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα απόβλητα ως ένα πόρο, αυτό είναι μια σημαντική στρατηγική, αλλά είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και από πριν ποια είναι τα υλικά τα οποία θέλουμε να βάλουμε στην οικονομία, η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τη μεγιστοποίηση των πόρων που ανακυκλώνονται και έτσι να σταματήσουμε και να, ή να μειώσουμε τουλάχιστον την εξάρτησή μας από πεπερασμένους πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Πέτερ Κούρθ που είναι από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διαχείρισης ε, Αποβλήτων και Υπηρεσιών για το Περιβάλλον. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ένα διαδικαστικό. Δεν έχουμε αντίτυπα των παρουσιάσεων. Δεν είναι διαθέσιμα στο e-committee, δεν τα βρίσκω πουθενά και είναι λίγο δύσκολο να διακρίνουμε την οθόνη από εδώ. Υπάρχει τίποτε διαθέσιμο. Πρόεδρος, θα ρωτήσω. Okay. Uh, ναι. Ευθύς αμέσως θα λάβετε αντίτυπο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, βουλευτές θέλω να σας ε, ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση αυτή και την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την οργάνωσή μας για τη διαχείριση των ε, αποβλήτων. Εμείς εκπροσωπούμε τις οργανώσεις από ε, τα 18 κρατη και επίσης τη Σερβία και την <clears throat> Νορβηγία και έχουμε ένα πολύ ψηλό κύκλο εργασιών. Ο κ. Ποτότσνικ είχε πριν από δύο χρόνια παρουσιάσει αυτό το πακέτο και ε, η απόσυρσή του σε πολλές απόψεις ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι λαθασμένο. Υπήρξαν βέβαια ορισμένα σημεία τα οποία ήταν προς βελτίωση στο πακέτο αυτό. Και αυτό έχει να κάνει και με την νομοθετική διαδικασία. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι λαθασμένο μήνυμα το να διακοπεί η νομοθετική διαδικασία και να αποσυρθεί η πρόταση αυτή. Για μένα θα ήταν πιο σημαντικό να δώσουμε έμφαση στους σωστούς στόχους και τις ε, μεθόδους που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές για την κυκλική οικονομία του αύριο. Ξέρουμε όλοι ότι στο παρελθόν τα μέσα τα οποία τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την Κομισιόν δεν χρησιμοποιήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν για την ε, βελτίωση χωματερών και δεν δημιούργησαν σε κανένα βαθμό την απαραίτητη υποδομή για μια κυκλική οικονομία. Υπάρχει μια ιεραρχία για τα απόβλητα που προβλέπεται από την αρμόδια ε, οδηγία και μπορούν εδώ να υπάρξουν σημαντικές πρόοδοι με μια εταιρική σχέση τομέα. Είναι απαραίτητο όμω να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για τη δημιουργία ενό νομοθετικού πλαισίου, αλλά κυρίω σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τα απόβλητα, το οποίο να καλύπτει όλη την Ευρώπη και το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση σε μια υποδομή για την αντιμετώπιση των αποβλήτων που αντιμετωπίζει σωστά την ιεραρχία των αποβλήτων. Παραδείγματο χάρη, η επιλογή, η διαλογή μάλλον των τεχνητών υλικών θα πρέπει να εξασφαλίσει την ε, επιλογή από απόβλητα η οποία απαιτεί ένα, μια κρίσιμη μάζα που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια άτομα. Υπάρχει η γενική άποψη πρέπει να κινηθούμε προς μια πιο οικολογική βιομηχανική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι μπορούν να δημιουργηθούν πάνω από 500.000 θέσεις στον τομέα αυτό. Στη Γερμανία ήδη 250.000 και παραπάνω άτομα εργάζονται στον τομέα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία αναφέρει η Κομισιόν είναι εφικτά. Η μείωση των αερίων θερμοκηπίου και η καλύτερη χρήση των ε, εναλλακτικών ενεργειών μπορούν να μας δώσουν περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και επομένως το ρόλο αυτό που μπορούν να παίξουν οι πρωτοβουλίες αυτές που παρουσιάζουμε σήμερα δεν πρέπει να τον παραγνωρίσουμε. Ένα σημαντικό τμήμα αυτού του πακέτου για τα απόβλητα φαίνεται και από τις δομές οι οποίες δημιουργούνται χώρες όπως η Σκανδιναβία, το Βέλγιο, η Γερμανία δεν θα έχουν μεγάλες δυσκολίες. Αλλά είναι πολλές οι χώρες οι οποίες θα έχουν δυσκολία για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης 50% ανακύκλωσης. Και για τις χώρες αυτές η απόσυρση του πακέτου δείχνει ότι σε περίπτωση δυσκολιών ε, μπορεί κανείς να αγνοεί την κατεύθυνση αυτή που δίνει η Ευρώπη. Σας παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε και πάλι και να μην δώσετε ένα τέτοιο λανθασμένο μήνυμα. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Πιότρ Μπέρθακ, υπεύθυνο για τα απόβλητα στο Ευρωπαϊκό ε, Περιβαλλοντικό Οργανισμό. Ευχαριστώ. Ε, δουλεύω για το ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση. Βλέπουμε ποια είναι η επίδραση του χώρου των αποβλήτων ε, στην πρόταση για την κυκλική οικονομία και βλέπουμε τι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα θέματα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα κινηθούμε για να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων και να μοιραστούμε τις ε, σωστές εμπειρίες μεταξύ μας. Είμαστε μια ομοσπονδία μη κυβερνητικών οργανώσεων με 50 εκατομμύρια πολίτες ως μέλη μας. Στις Βρυξέλλες είμαστε ένα συνασπισμός με κυβερνητικών οργανώσεων και θα παρακαλούσα να κοιτάξετε τις δηλώσεις τους εδώ. Ανατρέπονται με τα όσα αναφέρονται εδώ όλα τα ψευδεπιχειρήματα του κυρίου Τίμερμανς, τα οποία όχι μόνο δεν ευσταθούν, αλλά μπορούν και να ανατραπούν. Βλέπετε στο έγγραφο τι γίνεται με, τα, με τους περιορισμούς που υπάρχουν στον πλανήτη μας ε, με την ε, δυνατότητα απορρόφησης των αποβλήτων. Αυτό που θέλουμε είναι ευημερία στα όρια του πλανήτη. Η πρόταση για τα απόβλητα είναι ως τώρα το μόνο πρακτικό εργαλείο που έχουμε για να πετύχουμε τους δεσμευτικούς στόχους που έχουν προβλεφθεί όπως ο στόχος υπαριθμών 2 για την ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων ή τον τρίτο. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν καθυστερήσεων, διότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δάλλως δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας ως το 2020. Να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που στήριξαν με τις ψήφους τους την περασμένη Πέμπτη που στήριξαν την διαφωνία με την απόσυρση της πρότασης από το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής. Βλέπετε ότι τρεις από τις τροπολογίες που αφορούσαν το θέμα αυτό ψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Ακόμη και αν δεν υπήρχε ψήφισμα που έχει μια πολιτική βαρύτητα, υπήρξε ένα σαφές μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κοφεύει σε τέτοιες προτάσεις. Βλέπετε και επιστολές των Ευρωβουλευτών που το αποδεικνύουν. Και ακόμη και αν τον ε, Οκτώβριο παρά τους ενδιασμούς τους τα κάτι μέλη καλωσόρισαν το πακέτο, το επανέλαβαν το Δεκέμβριο με το Συμβούλιο. Καλωσορίστηκε το πακέτο στην τωρινή του μορφή, δηλαδή είναι αντίθετη με την απόσυρση του πακέτου. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών επίσης εργάστηκαν επί του θέματος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δημοτικές αρχές, η βιομηχανία, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλες οι φωνές αυτές αγνοήθηκαν από τον Επίτροπο Τίμερμαντς. Νομίζω ότι πρέπει να εξώσουμε το ανάστημά μας και να διαμαρτυρηθούμε. Ας περάσουμε τώρα στην ουσία. Βλέπετε πόσο έχει γίνει της μόδας η κυκλική οικονομία θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά να πω ότι το πλεόνασμα που αναφέρεται εδώ δεν έχει σκοπό να συγκεντρωθεί γρήγορα. Δηλαδή ο κύκλος ζωής των προϊόντων πρέπει να παραταθεί με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης μικροί όγκοι. Γιατί, γιατί όπως είπα, οι ροές των αποβλήτων δεν είναι ενδεικτικέ αναγκαστικά. Πρέπει να αποφύγουμε κάθε περιττό απόβλητο, όπω μοναδικής τα ε, μοναδική χρήση αντικείμενα. Τώρα, μία ερώτηση. Πώ να ξαναφέρουμε το βιομηχανικό αυτό κλάδο πίσω στην Ευρώπη. Καλή σα τύχη αν προσπαθήσετε, αλλά νομίζω το καλύτερο είναι να δώσουμε κίνητρα στην βιομηχανία μετά την κατανάλωση, δηλαδή τις ε, δράσεις επισκευής και ανακύκλωσης. Αυτές τις δραστηριότητες μπορούμε να τις ξαναφέρουμε στην Ευρώπη. Και αυτό ισχύει για τα ηλεκτρονικά, τα κλωστοϋφαντουργικά, τα πλαστικά και ούτω καθεξής. Έχουμε ετοιμάσει μια έκθεση που μπορείτε να την κατεβάσετε και από τον ιστότοπό μας και εκεί αναφέρουμε ότι πάρω από 800.000 θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τον βιομηχανικό αυτό κλάδο. Δηλαδή ένα στου έξι ανέργου θα ξαναβρούν δουλειά, ιδίω μεταξύ των νέων. Τώρα, στην αποτέφρωση, πόσε θέσει εργασία. Αυτό είναι μια ερώτηση προ εσά. Να πω ότι είναι σημαντικό να έχουμε δεσμευτικούς στόχους. Το τονίζω. Γιατί αριστερά βλέπετε την ανακύκλωση υλικών. Σε μια δεκαετία έχουμε προχωρήσει. Γιατί, Γιατί είχαμε δεσμευτικούς χρο... Ε, στόχους. Με τα ε, οργανικά απόβλητα, τα βιολικά απόβλητα όμως βλέπετε ότι δεν, υπήρξαν, δεν υπήρξε πρόοδος γιατί δεν υπήρχαν δεσμευτικοί στόχοι. Έχουμε και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη της Ευρώπης που θα μας απασχολήσει ως θέμα πολύ τους ερχόμενους μήνες. Το είπε και ο συνάδελφος. Χρειαζόμαστε νομοθεσία που ανακαλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι πρόεδρο τη ομάδα για τα απόβλητα, όπου συγκεντρώνονται οι πυρογνώμονε περί αποβλήτων από όλη την Ευρώπη, Ανατολική, Κεντρική. Και είμαι Πολωνό. Ξέρω την κατάσταση τη Τσεχία και τη Σλοβακία πολύ καλά. Τα σχέδια διαχείριση των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί από του υπουργού περιβάλλοντο εκεί δεν είναι καθόλου φιλόδοξα. Το ίδιο το σύνθημα το ακούμε και από του πολιτικού μα. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά μέτρα. Οι χώρες από μόνες τους δεν θα κάνουν τίποτα. Το έχουμε δει αυτό από την ιστορία ως τώρα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένους υπολογισμούς, ε, οικολογικό σχεδιασμό και πολλά ακόμα που δεν έχω χρόνο να τα αναπτύξω. Συμπέρασμα. Τι σημαίνει να έχουμε φιλοδοξότερη πρόταση αφού αποσύρθηκε. Για μένα και τους συναδέλφους με τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις μία λύση υπάρχει. Να μείνουμε στο ίδιο επίπεδο φιλοδοξιών και να διατηρήσουμε τις καλές πρωτοβουλίες που έχουν συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση για την κυκλική οικονομία. Με εισηγήτρια την κυρία Πιτικάινεν. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στο νομοθετικό τμήμα της πρότασης. Αυτό θα ήταν το πιο φιλόδοξο και δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε τίποτε άλλο. Ολοκληρώνω στο δυνατόν συντομότερα. Το μέλλον της Ευρώπης θα ήταν πιο φωτεινό. Έχουμε όλο τα υλικά και μας λείπει ο διακόπτης και η πολιτική βούληση. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μπραντολίνη, μέλος της Ευρώπης των Δημοτικών Αποβλήτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσκληση να πω ότι εκπροσωπώ δύο ευρωπαϊκές ενώσεις, την Ευρώπη των Δημοτικών Αποβλήτων, που ε, συγκεντρώνει μια ομάδα φορέων που διαχειρίζονται απόβλητα και επίσης την ε, CEP που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο των Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες με παρουσία πολλών ε, μελών μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δύο αυτοί φορείς, η CEP και η MWE, έχουν καλωσορίσει το πακέτο για την κυκλική οικονομία ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για μια κυκλικότερη οικονομία ε, με αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Αυτό θα είναι μια κινητήριος δύναμη και για την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορθώς το πακέτο για την κυκλική οικονομία εντοπίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η διαχείριση αποβλήτων. Ως ε, διαχείριση αποβλήτων εννοούμε την ε, ορθολογιστική, την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ε, να τονίσουμε ότι για την πλήρη υλοποίηση της ορθολογιστικής χρήσης αποβλήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας πρέπει να ξεκινήσουμε από την πρόληψη και την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση. Ε, βήματα καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία όλου του πακέτου. Το πακέτο για την κυκλική οικονομία προτείνει να διατηρηθεί και μπορούμε να το συζητήσουμε ως προς το περιεχόμενο. Το πακέτο λοιπόν έλεγα για την κυκλική οικονομία μας προτείνει ένα νέο ορισμό των δημοτικών αποβλήτων. Θεωρούμε ότι ο ορισμός αυτός μπορεί αποκλειστικός να συμφωνεί με την προέλευση, τη φύση και τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση των ίδιων των αποβλήτων. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με συμφέροντα εταιριών ή κοινοτήτων που παράγουν απόβλητα ή την ε, με τη συλλογή αποβλήτων. Θεωρούμε, ε, θεωρούμε ότι οι στόχοι της ανακύκλωσης είναι σημαντικοί στόχοι και υπάρχει ανάγκη για ενιαία, ομοιόμορφη μέθοδο σε επίπεδο κρατών μελών για να υπολογίσουμε το ποσοστό ανακύκλωσης. Θεωρούμε ότι η μέθοδος υπολογισμού πρέπει να βασιστεί στα πρώτα αποτελέσματα της επιλογής που θα γίνει. Επίσης ε, εντοπίζουμε την ανάγκη να υπάρξουν δεσμευτικοί φιλόδοξοι στόχοι. Αλλά οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Και ε, να μπορεί κανείς να τους ε, επιτύχει. Οι νέοι στόχοι θα πρέπει ως εκ τούτου να σχεδιαστούν καταλήλως, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο. Το πλαίσιο που μας αναγκάζει να ορίσουμε με διαφορετικό τρόπο τα δημοτικά απόβλητα και νέες μεθόδους υπολογισμού αλλά και την ανάγκη να έχουμε μια συνειδητή καταγραφή των αποτελεσμάτων από τη διαχείριση των αποβλήτων, που τώρα δεν καταγράφονται παρκώς σε 28 τουλάχιστον χώρες. Πιστεύουμε επίσης ότι η ανακύκλωση πρέπει να ενταθεί, ε, να ε, γίνει περισσότερο διαδεδομένη και ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα, ώστε να υπάρχει ανακύκλωση των υλικών. Επίσης πρέπει να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι ανακύκλωσης για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων, ιδιαιτέρως για, για τα πιο σημαντικά, όπως τα τροφικά αποβλήτα και τα βιολογικά. Θεωρούμε ότι η εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού είναι σημαντικό εργαλείο για να επιδιώξουμε τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και για να υπάρξει αποτελεσματικότερη και πιο επιτυχημένη επιδίωξη των υψηλότερων στόχων ανακύκλωσης. Να προσθέσουμε ότι η αγορά των ανακυκλωμένων υλικών πρέπει να ενδυναμωθεί. Υπό αυτήν την έννοια η κατάρτιση κριτηρίων για το τέλος των αποβλήτων θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως σημαντική ευκαιρία. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι ο οικολογικός σχεδιασμός θα είναι το κλειδί που θα μας ανοίξει την πόρτα στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους εφόσον είναι και επιτεύξιμοι στα θέματα της ανακύκλωσης. Οι στόχοι της ανακύκλωσης θα πρέπει να συνοδευτούν από μια αξιοποίηση των υποδομών που υπάρχουν για την ανακύκλωση, αλλά υπάρχει ανάγκη να σχεδιαστούν και για λόγους βιομηχανικής ανάπτυξης σχέδια διαλογής και επεξεργασίας των βιολογικών αποβλήτων. Αυτό, όπως έχουν δείξει ως τώρα παραδείγματα που έχουν ολοκληρωθεί σε πολλά κράτη-μέλη, αυτό είναι και μια σημαντική ευκαιρία για να υπάρξει ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στις χώρες μας. Οι επιδόσεις των κρατών μελών στην ε, διαχείριση των αποβλήτων δείχνει ότι παραμένει η ανάγκη να αναπτυχθούν τέτοιου είδου υποδομέ. Ιδίω για την ανακύκλωση και την ε, ανάκτηση. Και κάποιες σκέψεις για τους στόχους. Τους ε, στόχους της αποκομιδής και των ε, χήτα. Οι στόχοι όπως συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, ένα τρόπος επιδίωξη της κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστέ να προχωρήσουμε σταδιακά με μικρά ρεαλιστικά βήματα. Τα steps, τα βήματα που έχουν καθοριστεί στο 2025 και 2030 είναι νομίζουμε κατάλληλα. Οι στόχοι της αποτέφρωσης, όπως και οι στόχοι της ανακύκλωσης, θα πρέπει να ισχύσουν για όλα τα απόβλητα και όχι μόνο για τα δημοτικά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε και τώρα τελευταία παρέμβαση πριν περάσουμε στη συζήτηση η Βιρτζίνια Γέντσεν, εκτελεστική διευθύντρια της European. Παρακαλώ. Θα να σας ευχαριστήσω προσκαλέσατε τη Europen στη σημερινή ακρόαση. Θέλω να ευχαριστήσω τους και εισηγητές και τους αξιότιμους βουλευτές που παρευρίσκονται στην ακρόαση. Η πλειοψηφία των βουλευτών έχουν υποστηρίξει το τωρινό πακέτο για τα απόβλητα και ελπίζω να είναι σημαντική έκφραση αυτής της υποστήριξης σημερινή ακρόαση, όπως είπε και η κυρία Μποναφέ. Εξ αρχής υποστηρίξε η Europen το πακέτο και ζήτησε βελτίωση για τρία βασικά σημεία που θα σας περιγράψω. Θα συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε, ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το στόχο για την κυκλική οικονομία. Europe είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συσκευασία και για το περιβάλλον. Ε, λίγο ασυνήθιστη ένωση, εκπροσωπούμε εξορροπημένες απόψεις από ολόκληρη την αλυσίδα. Ε, παραγωγή, ε, παραγωγή των συσκευασιών, χρήση χρήστες ε, δεν ε, ε, υπάρχει κάποια προτίμηση για τα υλικά συσκευασία. Σε πάνω από 20 χρόνια συνεργαζόμαστε τόσο ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα τη συσκευασία. Χρειαζόμαστε μια δαιμονισμένη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσουν να λειτουργούν επιχειρήσει, να είναι ανταγωνιστικέ και να βρίσκουν καινοτόμε λύσει που καλύπτουν τι περιβαλλοντικέ αλλά και τι οικονομικέ συνιστώσει μπορούμε με ένα εφικτό, θεμητό και εναρμονισμένο πλαίσιο να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και σας είπα ότι υπάρχουν τρεις βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν κατά τη γνώμη μας. Πρώτον, εναρμονισμένοι ορισμοί και οι ρεαλιστικοί στόχοι για την ανακύκλωση. Δεύτερον, να προσδιορίσουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε αυτό συμπεριλαμβανομένης και της εκτεταμένης ευθύνης των παραγωγών υλικών συσκευασία και τρίτον, αγορά, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων συσκευασία ε, θα πρέπει να παραμείνει μια θεμελιώδης αρχή στη νέα οδηγία για τα απόβλητα και τα απόβλητα των συσκευασιών. Χρειαζόμαστε καινοτομία, νέες τεχνολογίες και έτσι μόνο θα κατοχυρωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα λεπτά που μου απομένουν για τρία βασικά μήνυματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση μέτρησης, δηλαδή να έχουμε αρμονισμένους ορισμούς ε, που θα χρησιμοποιούμε για την μέτρηση ε, των συσκευασιών και αυτό να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους που θα βασίζονται στους αρμονισμένους ορισμούς, δηλαδή δηλαδή στο πρώτο βήμα. Γιατί ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει γι' αυτό, διότι αυτή είναι η βάση για να υπάρξει μια ε, χρήστη πολιτική διαχείριση των αποβλήνων και να γίνουν οι απαιτούμενε επενδύσει. Ε, υπάρχουν πολύ μεγάλε προκλήσει στι οποίε θα πρέπει να αντεπεξέλθουμε για να υλοποιήσουμε όλου του υπόλοιπου στόχου ε, στην πολιτική αποβλήτων. Η νομοθεσία στα κράτη-μέλη διαφέρει σημαντικά και λόγω αυτών των σημαντικών διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν, μα εμποδίζουν από να υλοποιήσουμε του στόχου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποδομέ για τη διαχείριση των αποβλήτων, επίπεδα αποδοτικότητα, σε τέτοιε παραμέτρε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν θέτουμε του νέου στόχου. Μετά τη μέτρηση, την εναρμονισμένη μέτρηση, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα υλοποιήσουμε αυτού του στόχου. Και φτάνουμε στο EPR, την εκτεταμένη ευθύνη παραγωγού, δηλαδή ε, σε ένα πρώτο επίπεδο βλέπουμε την ε, επιχειρησιακή ευθύνη του παραγωγού, η οποία παρατείνεται μέχρι το τέλος ζωής του προϊόντος, μέχρι δηλαδή να υλοποιηθούν οι στόχοι. Τα συστήματα EPR λοιπόν έχουν δημιουργηθεί ούτως ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν ε, να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσει ε, για να ε, παραμείνει ένα επιτυχές εργαλείο το EPR θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει για τις επιδόσεις για το EPR μέσα στην οδηγία για τα απόβλητα και τα απόβλητα συσκευασιών. Έτσι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, στη διαχείριση δηλαδή των αποβλήτων συσκευασίας να έχουν το δικό τους ρόλο και βάσει της αρχής επικουρικότητας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραμένουν ε, ε, ελεύθερα ώστε να έχουν την απαιτούμενη ευελιξία στον προσδιορισμό των συστημάτων EPR για να ανταποκρίνεται αυτό στις τοπικές ανάγκες. Με τις ελάχιστες όμως απαιτήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσουμε ότι όλα τα συστήματα EPR, τα μη κερδοφορά για τους παραγωγούς και τα υπόλοιπα που δεν χειρίζονται πλέον οι παραγωγοί θα λειτουργούν βάσει των ίδιων αρχών και τα διάφορα μοντέλα EPR μπορούν να συνεπάρξουν με αυτόν τον τρόπο έτσι ε, η ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα και η καινοτομία θα τονωθούν και η διαφορετική ε, συλλογή και ε, διαχείριση των αποβλήτων ε, θα καταστεί δυνατή. Χρειάζεται όμως σαφήνεια ως προς το ρόλο και τις αρμοδιότητες σε κάθε οικονομικού φορέα για την εφαρμογή οποιοδήποτε συστήματος EPR. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία για όλους, για τις, τους παραγωγούς, για τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, για τους καταναλωτές, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα συστήματα EPR. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη σε σχέση με το ε, σε ποιον μπορούν να αποδοθούν οι ευθύνε και πού αρχίζει και πού τελειώνει η εκτεταμένη ε, ευθύνη για τον παραγωγό. Βάσει τωρινής πρότασης, ε, το συνολικό κόστο για την διαχείριση βαραίνει μόνο τον παραγωγό και δεν εξετάζεται ο ρόλο όλων των υπολείπων φορέων. Δηλαδή είναι λευκή επιταγή που μα επιβάλλεται και δεν έχουμε κανένα έλεγχο για την αποτελεσματικότητα και για τι επιδόσεις αυτών των συστημάτων EPR. Δεν έχω άλλο χρόνο για να σας μιλήσω μιλήσω για τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στη νέα νομοθεσία. Υπάρχει όμως ενημερωτικό δελτίο fact για το EPR και θα το βρείτε βγαίνοντας από την αίθουσα. Υπάρχει και το έγγραφο θέση μας για την ε, ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξίσου σημαντικό είναι το τελευταίο σημείο είναι η αρχή της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να παραμείνει η ραχοκαλιά της νέας οδηγίας για τα απόλυτα και τα απόλυτα συσκευασίων. Οικονομία κλίμακος, ισχυρότερος ανταγωνισμός, χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης, καλύτερη κατανομή ε, των πόρων, αυξημένη η επιλογή των καταναλωτών και ε, αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Να μην ξεχνάμε ότι ο λόγος ύπαρξης της οδηγίας αυτός ήταν όταν εγκρίθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 90, διότι η διαφορετική περιβαλλοντική κανόνες αν σε στρέβλωση και κολλήματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πορευμάτων και των συσκευασιών. Θα πρέπει να προστατευτεί η ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς ε, όμως ε, αυτό δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία ε, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιβάλλει στα κράτη-μέλη τι είδους νομοθεσία θα έπρεπε να υιοθετήσουν. Όχι, γιατί αυτό συνεπάγεται προστατευτισμό και κατάτμιση της εσωτερικής αγοράς υπονομεύοντας ε, τον ανταγωνισμό, την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας, υποσκάπτοντας έτσι την βασική επιταγή της κυκλικής οικονομίας. Ευχαριστούμε. Κλείνοντας θα ήθελα ε, μόνο να δούμε τα βασικότερα σημεία. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεισνομεθετική διαδικασία. Θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία. Λαμβάνουμε γνώστο ότι θέλει ε, να αποσύρει την πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταθέσει μια νέα πρόταση. Θα ε, συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία με εσάς και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τόσο ώστε η μελλοντική συνενομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει σαφής και να είναι ο κινητήριος μοχλός για οικονομική ανάπτυξη και να είναι κάτι το ρεαλιστικό. Σας ευχαριστούμε. Θα αρχίσουμε τώρα ευθύς αμέσως με τις ε, ερωτήσεις ε, των ε, σκιωδών και των μελών της Επιτροπής. Θα αρχίσω δώντας το λόγο στην κυρία Μποναφέ για να αρχίσει η συζήτηση. Ευθύς αμέσως να περάσω σε ερώτηση από ό,τι κατάλαβα, μπορούμε να πούμε και από την προηγούμενη συζήτηση ότι η μόνη αποδεκτή οτιολόγηση της πρότασης ε, που ακούσαμε από τον Διευθυντή Φάλκενμπεργκ είναι ότι λείπει ένα ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στο πώς να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές που πρέπει να μας οδηγήσουν στην επίτευξη των ε, φιλόδοξων στόχων για την ανακύκλωση. Ένα από του εισηγητές μα μίλησε για τα διευθυντικά ταμεία, όμω πέραν των διευθυντικών γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το επενδυτικό πρόγραμμα του κ. Γιούγκερ στη διάθεσή μα. Οπότε διερωτώ με, και το ρωτώ και προ τους εισηγητές, ε, τους μα, μας, πώς πιστεύετε ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βελτιωθεί για να πλησιάσουμε τους στόχου της ανακύκλωσης και την επίτευξή τους. Πρόεδρος, άλλες ερωτήσεις. Γιάννη. Το ίδιο ερώτημα ακριβώ είχα. Οπότε απλώ θέλω να ακούσω τι απαντήσει των ε, εμπειρογνωμόνων μα. Εντάξει. Άλλα ερωτήματα από τα μέλη μα. Όχι. Εντάξει. Ξεκινάμε από τον πρώτο μιλητή για να ακούσουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ετέθηκαν από την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν επενδύσεις για μένα σε συστήματα και υποδομές που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αντιμετώπιση των αποβλήτων, η συλλογή τους και η αντιμετώπιση τους ένα ουσιαστικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας να ξαναμπούν σε παραγωγικές ιδιαιτησίες τα, ε, σε παραγωγικές διαδικασίες τα υλικά αυτά και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για την ανάστροφη αυτή επιμελητία συλλογής των ε, προϊόντων. Πρέπει επίση και η βιομηχανία να επενδύει περισσότερο σε μια λογική από διάσπασης των προϊόντων που παράγει και να μην παράγει προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να αποσυνδεθούν μετά το τέλος της ζωής τους και ώστε τα υλικά αυτά να ξαναγυρίσουν σε παραγωγικές διαδικασίες. Τα συστήματα λοιπόν συλλογής και η ανάστροφη επιμελητία υπάρχει μεγάλο δυναμικό εδώ να εξετάσουμε τις ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν για τα υλικά που είναι παραγωγικά χάρη βιοαποδομήσιμα και να προωθήσουμε αυτή την πλευρά της οικονομίας σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, νέα υλικά που μπορούν να προκύψουν, τα οποία μπορούν να μπουν μέσα στο κύκλο παραγωγής, ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στο οικοσύστημα ή αλλιώς να διατηρηθούν μέσα στην, στο παραγωγικό βρόχο, γιατί κάποια από αυτά τα πρώτα υλικά μπορούν να ε, αντικαταστήσουν τα καινούρια να τα ήδη υφιστάμενα. Να έχουμε λοιπόν νέε μορφές σχεδιασμού και ανακύκλωση των υλικών μέσα στην ε, βιομηχανική παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ για το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια για το πώς τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μια τέτοια λογική και ιδίω αυτά τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν μια απαραίτητη υποδομή η οποία χρειάζεται για την ε, ανακύκλωση των υλικών. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι τα μέσα τα οποία ήταν διαθέσιμα από τις Βρυξέλλες δεν χρησιμοποιήθηκαν ή αλλιώς απορροφήθηκαν αλλά χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο ο οποίος δεν ήταν σύμμορφος με την οδηγία. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό έγινε η χρηματοδότηση αυτή για την ε, βελτίωση και την επέκταση ε, χωματερών, χήτα, και αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο προβλεπόταν με την ιεραρχία των αποβλήτων. Το Κοινοβούλιο είχε τονίσει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαφορετικά κονδύλια προς την κατεύθυνση αυτή για να υλοποιηθεί η ιεραρχία των αποβλήτων είναι σαφές ότι έχουν κατανοήσει ορισμένες χώρες ότι για τις πόλεις είναι απαραίτητο να υπάρξει μια δημιουργία των υποδομών για τα απόβλητα. Υπάρχει ακόμα το, το πρόβλημα όμω γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει κανείς χωματερές, είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει την υποδομή για αποτεφρωτήρες κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ε, πίεση ώστε όχι μόνο να χρησιμοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις αλλά να προσελκυθούν και επενδύσεις από το ιδιωτικό τομέα να γίνουν συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα γιατί θα πρέπει να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας μαζί με τις δημοτικές αρχές για να μπορεί να υπάρξει μια λύση για τα αστικά απόβλητα. Θέλουμε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο το υπόδειγμα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερο με αυτόν τον τρόπο, γιατί στο βαθμό που γίνεται όλο και πιο ακριβή η εναπόθεση σε χωματηρές, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρο να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις οι οποίες θα μειώσουν τον όγκο των υλικών που πηγαίνουν στις χωματερές. και από το νέο αυτό ταμείο μπορούμε να προσθέσουμε νέα κονδύλια και αν γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο αυτό θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη πρόοδος για τα νέα κυρίω να μπορέσει να υπάρξει αυτή η λογική ανακύκλωση. Α, για μένα λοιπόν φαίνεται <clears throat> να ε, είναι αντίφαση να θέλει κανείς να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και να αποσύρει από την άλλη μεριά μέτρα όπως αυτά για το νέο ταμείο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος γιατί τα εξήγησαν όλα πολύ ωραίοι συνάδελφοι. Πρέπει κυρίως στις ανατολικές χώρες ε, που έχουμε υστέρηση σε σχέση με την ανακύκλωση να προσέξουμε πάρα πολύ να μην επενδύσουμε σε ε, υπερβολικές ε, να μην επενδύσουμε με τρόπο ώστε να χάνουμε την ενέργεια. Ε, έχω την εντύπωση ότι το επενδυτικό σχέδιο Juncker θα ε, εφαρμοστεί ακόμη και αν ε, εξακολουθεί να ισχύει η τωρινή πρόταση της Επιτροπής για τα απόβλητα. Ίσως κάνω λάθος, αλλά θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε. Ο Δόκτωρ Μπαντολίνη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ερευνητική δραστηριότητα για τα θέματα αυτά, για τα υλικά και για τις παραγωγικές διαδικασίες για να εξασφαλίσει την ανάκτησή του στο τέλος της ε, ζωής ενός προϊόντος για να μπορέσει να, υπο, να υποστηριχθεί η ανακύκλωση και ακόμα και η παράταση της δυνατότητα χρησιμοποιήση αυτών των υλικών. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την έρευνα σε σχέση με συστήματα και διαδικασίες που θα επιτρέπουν να ανακτούμε και να ανακυκλώνουμε τα απόβλητα. Να βελτιώσουμε λοιπόν την αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων και επίσης να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ροές αποβλήτων που μέχρι στιγμής ξεφεύγουν από την προσοχή των ε, επιχειρήσεων και της κοινή γνώμη, αλλά όπου η ανάκτηση πόρων θα μπορούσε να είναι σημαντική, δηλαδή όλα αυτά τα απόβλητα να επαναχρησιμοποιούνται. Παραγωγή χάρη τα ύδατα καθαρισμού ή η, η, τέφρα των αποτεφρωτών. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να το πράξουμε αυτό, ιδίως στις περιοχές αυτές της Ευρώπης που έχουν τις ασθενέστερες υποδομές να μπορέσουν να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα συστήματα από τη στιγμή της συλλογής των αποβλήτων μέχρι τη στιγμή της ανάκτησης των ε, ε, υλικών που χρειάζονται ή μέχρι την τελική τους ε, εναπόθεση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν σχέδια για όλες αυτές τις περιοχές και θα πρέπει να προβλέψουμε να υπάρξουν εγκαταστάσεις για όλη τη φάση της ε, ανακύκλωσης που να συναρμόζονται με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Πιστεύω ότι πολλά καλά, ε, σωστές σκέψεις παρατηρήσεις είπαν οι προηγούμενες θα πρέπει να επενδύσουμε πρώτα απ' όλα ε, στην ε, διαφανή νομοθεσία για το θέμα των αποβλήτων. Ε, ήδη θα βοηθηθούν έτσι τα κράτη-μέλη που χρειάζονται υποστήριξη και ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων και όπως είπε και ο συνάδελφος θα πρέπει να επενδύσουμε σε καλύτερες πολιτικές συλλογής, των αποβλήτων, να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες, δυνατές, ε, βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές στα κράτη-μέλη. Φυσικά, για μας ήταν πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις στον καινοτόμο σχεδιασμό των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις ανάγκες των καταναλωτών ε, για να εξυπηρετεί το στόχο της συσκευασίας, συσκευασία, να είναι λειτουργική, οικολογική και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνονται επενδύσεις για την ε, ε, διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών για την καλύτερη διαλογή παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στα σχολεία γιατί είναι, ευκολότερη η διαπαιδαγώγηση όταν ε, ξεκινάει κανείς ε, από τις μικρές ηλικίε ε, για την διαλογή παραδείγματο χάρη. Πρέπει να σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι, κυρία Ποναφέ. Εγώ εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία αυτή για μια πιο ήπια ερώτηση. Μήπως αν θα πρέπει να υπάρξει και κάποια πτυχή για την ε, πρόληψη της ε, δημιουργίας αποβλήτων. Παραδείγματος χάρη υπάρχει αυτή η οδηγία για την ε, πρόληψη των αποβλήτων από τρόφιμα μέχρι το 2025 που πρέπει να εφαρμοστεί. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει ένα πιο φιλόδοξο βήμα στο πρώτο επίπεδο, το επίπεδο της πρόσληψης, πρόληψης των αποβλήτων. Έχουμε μιλήσει για αξιόπιστους στόχους. Θεωρείτε ότι τέτοιοι στόχοι για να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων μπορούν να είναι αξιόπιστοι. Ευχαριστώ. Και από τον κύριο Φλάνα ένα ερώτημα τώρα. Σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η η κυρία Γιάνσενς και για την καλύτερη εκπαίδευση των νέων και των ενηλίκων για την διαλογή των αποβλήτων. Αυτό πιστεύω ότι είναι εφικτό σε κάποιο επίπεδο, αλλά είναι τόσο πολλές οι ποικιλίε αποβλήτων που πρέπει να, διε, να, να Αυτό μπερδεύει πάρα πολύ κόσμο. Και όλα αυτά, <clears throat> εντάξει, μπορεί να είναι καλό για το περιβάλλον που λέμε ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας και να αφήνουμε το νερό να πιένσει στους υπονόμους και να παίρνουμε κάποιο υλικό και να το καθαρίζουμε με αυτόν τον τρόπο και μετά να το ανακυκλώνουμε. Ναι, καλά είναι αυτά, αλλά μήπως θα είχε περισσότερο νόημα να σταματήσουμε την έκπληση των υλικών για να μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε, να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα με πιο βιοαποδομήσιμα προϊόντα, τα οποία δεν χρειάζεται να πλένονται και με τον τρόπο αυτό μπορείτε να βάλετε περισσότερα υλικά σε ένα, ε, σε ένα καλάθι ή σε ένα κουτί, ώστε να μειώσετε την, ε, το μπέρδεμα της διαλογής. Και επίσης αυτό το οποίο ελέγχθη ήταν ότι θα ήταν πιο λογικό να μην αποσυρθεί το πακέτο για, την, ε, ε, για τα απόβλητα, αλλά να διορθωθεί. Αλλά ακόμα φαίνεται και ο τελευταίος επίτροπος δεν, το, δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτό το πακέτο. Και δίνω τώρα το λόγο για ένα τελευταίο γύρο στους εμπειρογνωμονές μας Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, για την αξιοπιστία και το εφικτό των στόχων από ποσοτικής πλευράς ε, ίσως δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο βήμα για να το συζητήσουμε αλλά θα συμφωνήσω με τον κύριο Φλάναγκαν που μόλις μας είπε ότι πρέπει να ανάντι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό είναι το μεγαλύτερο επόμενο βήμα και όχι να ε, ασχολούμαστε με πολιτικές ε, μετριασμού των ζημιών που αναγκαίες βέβαια είναι στη μεταβατική και Όντως πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, αλλά δεν φτάνουν. Μην ξεχνάμε ποιος είναι ο τελικός στόχος να σχεδιάζουμε τα απόβλητα τόσο ώστε στην τελική τους φάση να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα και όχι να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στο το, όταν προκύπτει και οι πολλήματα που δεν μπορούν να κυκλωθούν θα υπάρχουν πάντοτε. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά αν υπάρχει καλύτερο σχεδιασμό θα κλείσουμε τις τρύπες που υπάρχουν και θα έχουμε λιγότερα απόβλητα. νομίζω αυτό είναι το βασικό μήνυμα της κυκλικής οικονομία. Ο Υπάρχουν ακριβώς πώς πολλές έρευνες για το πώς γίνεται η διαλογή των αποβλήτων σαν, ε, με παράμετρο την ηλικία των ε, ε, καταναλωτών κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και τη διαδικασία που χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές καλές πρωτοβουλίες και ιδίως στον τομέα της ε, οικονομίας των παραγωγών να γίνεται η παραγωγή με καλύτερη εκμετάλλευση των πρώτων υλών και με λιγότερη παραγωγή ε, με λιγότερη κατανάλωση πόρων αλλά είναι δύσκολο να υπάρξει βελτίωση στα αστικά απόβλητα, στις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας χάρη, με τον γυράσκοντα πληθυσμό, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ένα δεύτερο ερώτημα για την ποιότητα της ε, ανακύκλωσης αυτή εξαρτάται από το να γίνεται έγκαιρα μια καλή, ένας καλός διαχωρισμός των αποβλήτων. Μπορούμε, γίνεται σωστά η διαλογή ήδη ε, στη, στα νοικοκυριά και αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το αποδέχονται οι πολίτες και οι καταναλωτές. Και εάν μπορούμε να βελτιώσουμε την διαλογή στο πρώτο επίπεδο, θα είναι πολύ καλύτερα από κάτι που γίνεται σε ένα αργότερο επίπεδο που δεν νομίζω μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστώ για αυτό το καλό ερώτημα για την ε, μείωση. Ε, και το πώ θα πετύχουμε τους στόχους. Ε, Όντω, πρέπει να το δούμε στο εγγύ μέλλον πριν την έγκριση. Αλλά όταν μιλάμε για την πρόληψη και έναν μόνο στόχο να προτείνεται, ούτε καν δεσμευτικό για τα τροφικά απόλυτα, 30% είναι πολύ μετριοπαθή στόχος. Εμεί θα θέλαμε 60%. Είμαστε φιλόδοξοι προ αυτό. 30 είναι απολύτως εφικτό. Εάν δείτε την ε, παραγωγή αλυσίδα των τροφικών αποβλήτων, όχι μόνο τα εργοστάσια, αλλά και το τι γίνεται με τους καταναλωτές, η βιώσιμη γεωργία και η προμήθευση είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Από το Γενικό Γραμματέα βεβαίως, ε, παρόλο που είχε ετοιμαστεί από τον κύριο Ποτόσνικ, ε, εμποδίστηκε ένα έγγραφο για, τη, για τα τροφικά απόβλητα. Είναι σημαντικό να δούμε την τροφική αλυσίδα λοιπόν και την μείωση που μπορούμε να πετύχουμε εκεί. Θεωρούμε πάνω απ' όλα ότι όταν ε, μιλά κανείς για πρόληψη ουσιαστικά εννοεί την ε, ορθολογιστική χρήση των πόρων. Θεωρούμε ότι εκπροσωπώντας τους ε, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή όταν τα απόβλητα έχουν φτάσει πλέον να είναι σε αυτή τη μορφή, πρόληψη θα πει αποτελεσματική χρήση των πόρων αλλά και του κύκλου των αποβλήτων. Διότι αν παράγουμε απόβλητα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, θα πρέπει να βρούμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά, τα συστήματα αποκομιδής, τα συστήματα διαχείρισης, δηλαδή τους οικονομικούς πόρους που χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση των ε, αποβλήτων για την πρόληψη Φαίνεται να υπάρχουν πολλές θεωρητικές δηλώσεις, αλλά οι πράξεις έλειψαν. Ήταν δηλές πρόληψη. Σημαίνει να εργαστούμε ως προς τον οικολογικό σχεδιασμό, να καθορίσουμε κανόνες σημαντικούς και φιλόδοξους για την ευθύνη, την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού σε σημείο που να μπορέσουμε να χαράξουμε σωστότερους στόχους. Να υπογραμμίσω ότι στη χώρα μου, την Ιταλία, εδώ και κάποια χρόνια, με την ε, οικονομική κρίση υπήρξε σημαντική μείωση παραγωγής αποβλήτων. Δεν ήταν βέβαια αποτέλεσμα ενάρετης προσπάθειας, αλλά ήταν ε, άμεση αποπτώση της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά υπήρξε αποσύνδεση αντίστροφη, αν μπορώ να το πω έτσι. δεν ε, ενισχύθηκε το ΑΕΠ από την ε, μείωση αποκομιδής. Ακόμη όμως δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι εφικτοί όπως είπα εφικτή εφόσον συνειδητά τους καθορίσουμε και τις απαραίτητες δράσεις που θα πρώτο συνοδεύουν. Η κυρία Γιάνσενς. Ευχαριστώ για την πρόληψη. Είναι σημαντικό και εξάλλου από επιχειρηματική ε, πλευρά ε, είναι πιο ενδιαφέρον να γίνεται η πρόληψη. Ε, ξέρετε ότι οι χρήστε δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε δεκάρα παραπάνω σε σχέση με τη συσκευασία που χρειαζόνται και για να βελτιωθούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τι συσκευασίε τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίση να ασχοληθούν εκείνα με το σχεδιασμό, ώστε να βοηθήσει αυτό ο σχεδιασμό για την πρόληψη για να μην έχουμε τόσο πολλά απόβλητα από τις συσκευασίες, απόλυτα τροφίμων κτλ. Ε, οι δυνάμεις της αγοράς ε, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένους στόχους, ε, αποδεδειγμένα είναι δύσκολο να γίνουν οι μετρήσεις ε, για να συλλέξουμε τα δεδομένα και γι' αυτό με να αναθεώρηση και την νομοθεσία σκοπούμε στις αυξημένες επενδύσεις για την ανακύκλωση και ε, την στήχηση των ε, στόχων ε, ανακύκλωσης με μια βάση για την μέτρηση με νέες νομοθετικές διατάξεις, να έχει ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο για την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού, ούτω ώστε όντως να υπάρχει καλύτερη διαλογή για τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και για τη συλλογή τους, να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης, γιατί και αυτό είναι μέτρο που χρειαζόμαστε για την πρόληψη. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε εγκαίρως. Λέω Πρόεδρος και νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ακρόαση ευχαριστώντας τους ε, εμπειρογνώμονες για τις παρεμβάσεις τους και για τη συμμετοχή τους. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου το απόγευμα και στις 29 έχουμε πρωί απόγευμα συνεδρίαση. Ευχαριστούμε. Καλή όρεξη.